Colleagues, good morning. Let's start our meeting. Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίασή μας. Έχω μερικές ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, να καλωσορίσω ένα νέο μέλο, Τον κύριο Σάντερ Λούνς, από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Θα αντικαταστήσει τον κύριο Φανόβερφελτ, ο οποίος, όπω ξέρετε, διορίστηκε Υπουργό Οικονομικών στο Βέλγιο. Καλώς ήρθε, Σάντερ. μετά έγκριση του σχεδίου χρονοδιαγράμματος για το 2015 με συνεδρίαση στις 13 όπως συμφωνήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τις ημερομηνίε των συνεδριάσεων και στο νηστότοπο τη επιτροπής. Επίση, αποφάσεις από την συνεδρίαση των συντονιστών. Πρώτα απ' όλα για το διορισμό των μελών του Συμβουλίου του SRM. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να οργανώσουν ακροάσεις για όλες τις ε, θέσεις του Συμβουλίου του SRM με βάση της νομοθεσίας και οι συνάδελφοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες των ακροάσεων εν ευθέτω χρόνο. Οι διορισμοί για τις εκθέσεις τώρα, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τις Οικονομικές Πολιτικές και το Συντονισμό τους, ΕΛΚ, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ρόλο του Διεθνούς ε, ε, Νομοθετικού πλαισίου και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ΑΛΔΕ, ε, έκθεση αντικτύπου για τι ε, χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε και την νομοθεσία του ΕΛΚ, έκθεση ιδέα πρωτοβουλία για τι επενδύσει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και η απόφαση απαλλαγή για τα ΕΖΑΣ από τα μέλη του Προεδρείου. Ενημέρωση τώρα για τη διαδικασία διορισμού για το ΕΣΚΑΠ. Ε, οι συντονιστές της Επιτροπής μας αποφάσισαν να γίνει ακρόαση με, τους τον υποψήφιο για την έδρα του ε, Συμβουλευτικού Συμβουλίου για τα στατιστικά στοιχεία. Θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία. Και τέλος, για την οικονομική διακυβέρνηση, οι συντονιστές της ε, Επιτροπής Οικονομικών θα διοργανώσουν οικονομικό διάλογο με τον Επίτροπο Μοσκοβισή στις 24 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο σε πρώτη φάση για να συζητήσουν τα σχέδια προπολογισμού των κρατών μελών. Σημείο 7. Πρέπει να ψηφίσουμε. Επανέρχομαι στην τελευταία μου ανακοίνωση. Ηλεκτρονική παρουσίαση για το e-committee, ε, παρουσίαση για το e-committee, ε, σύντομη παρουσίαση για την υπηρεσία αυτή του Κοινοβουλίου για την ηλεκτρονική συνεδρίαση, το e-meeting. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε το e-meeting εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Το e-meeting είναι μια εφαρμογή που σας παρέχει τα έγγραφα σε ηλεκτρική μορφή. Αντικαθιστά αυτά τα έγγραφα που λαμβάνετε σε χαρτί, σε φάκελο για τις συνεδριάσεις. Κάτι το οποίο ακόμα το έχετε, αλλά πρόκειται για μια ηλεκτρονική εκδοχή και έχει και γι' αυτό και άλλα ε, πλέον εκτίματα σε σχέση με το απλό χαρτί. Uh, uh, οπότε θα δείτε πώς λειτουργεί και θα δείτε και αυτά τα πλέον εκτίματα από αυτή μας την παρουσίαση. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε κατευθείαν θα σας κάνουμε αυτή την επίδειξη και η σκητάλη ανοίγει στον συνάδελφο. Καλημέρα σας λέει ο συνάδελφος. Οπότε έχουμε αυτή την εφαρμογή που είναι τέτοιου είδου που δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε τίποτα σε οποιοδήποτε συσκευή. Σήμερα να σας πούμε ε, τι ισχύει επί τη βάση του iPad, αλλά ισχύει και για, όλες τις άλλες, ε, για όλα τα άλλα tablets. Οπότε για να έχετε την πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε πάτε εδώ πέρα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ε, και μετά κάθετος e-meeting βάζετε στη συνέχεια και είναι εσωτερικού Δηλαδή είναι προσβάσιμη αυτή η εφαρμογή μόνο για τους υπαλλήλου, τους βουλευτές, τους συνεργάτες. Οπότε εδώ βάζετε αυτό το, το, το, το συνήθι κωδικό τον οποίο έχετε και τον κωδικό χρήστη βάζω το, το δικό μου. Once we in, we go directly to the... Οπότε κατευθείαν αυτό σας βγάζει στην ε, σελίδα τη βασική και βλέπετε ότι εδώ σας δίνει την δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε συνεδρίαση η οποία έχει ανέβει, έχει καταχωρηθεί εδώ. Οπότε εδώ έχετε μόνο τρία βήματα να κάνετε με το start, με την είσοδο αυτή. Είπαν πρέπει να είσαστε εδώ για να μπείτε στο e-meeting. Και, και εκτός κοινοβουλίου μπορείτε να έχετε πρόσβαση και δεν βλέπετε εδώ πέρα όλες τις επιτροπές να πάμε στη σημερινή μας συνεδρίαση. Βλέπετε εδώ πέρα όλ, ε, ενημερωμένα όλα τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν, όλες τις, ε, ε τις διατάξεις. Πάμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις, μπορούμε να δούμε και κάποιες μελλοντικές. Εδώ στα δεξιά μπορείτε να δείτε την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και μπορείτε εδώ πέρα να έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, όλα αυτά ηλεκτρονικά Βλέπετε εδώ πέρα όλες τις ε, υπάρχουσες γλωσσικές εκδοχές για κάθε έγγραφο. Επίσης, να ανοίξετε το έγγραφο στην τελευταία του εκδοχή. Αυτό το κατεβάζετε εδώ, το οποίο σημαίνει στην συσκευή την οποία και χρησιμοποιείτε. Να δούμε τώρα ένα άλλο έγγραφο, να το μπορώ να έχω πρόσβαση σε αυτό, μπορώ να το ανοίξω όμως και σε μια άλλη ε, συσκευή και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, να μπορώ να το επισημειώσω ας πούμε το έγγραφο, μπορώ να προσθέσω ένα σχόλιο Όλα αυτά τα οποία τα κάναμε στο χαρτί το οποίο χρησιμοποιούσαμε πριν και μόλις γίνει αυτό μπορούμε επίσης αυτό το έγγραφο να το στείλουμε σε έναν συνάδελφο με αυτές τις παρατηρήσεις, τις σημειώσεις που έχουμε γράψει. Και το e-meeting υπάρχει ανα πάσα στιγμή για, για όλες τις συνεδριάσεις. Μπορείτε να βρείτε και κάτι που έγινε πέρσι. Να μια σύντομη παρουσίαση. Η συναδελφός τώρα θα σας παρουσιάσει το e-committee. Καλημέρα. Λίγα λόγια για το e-committee και συγκεκριμένα το νέο site που έχουμε στήσει για την εξέταση των πράξεων εξουσιοδότηση και κατανάθεση. Μπαίνετε στο ίντρανετ, μπαίνετε μετά στο e-committee, μετά πάτε κάτω-κάτω εκεί που λέει Econ Workspace όταν το πατήσετε αυτό, κάντε ξανά login. Πρέπει να ξαναμπείτε γιατί το site ε, το οποίο έχουμε βάλει ε, είναι προσβάσιμο μόνο στα μέλη της Επιτροπής και του συμβούλους ε, των ομάδων. Μπαίνετε εκεί πέρα με τα γνωστά, το γνωστό όνομα χρήστη και συνθηματικό και μετά βλέπετε τον αυτό site που έχουμε για την εξέταση των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Εδώ πέρα βρίσκεται κατά βάση τέσσερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα μια εισαγωγή. Την δημιουργήσαμε μέσα Σεπτεμβρίου και στόχος είναι να αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες ε, για πράξη κατεξιοδότηση, για εφαρμοστικά μέτρα και όλα αυτά τα στέλνουμε με email σε ένα μέρος, στο site αυτό, για την ώρα. Το επόμενο που βλέπετε είναι τα τρέχοντα ζητήματα όλα όσα έχουμε δώσει δηλαδή στα μέλη της ΕΚΟΝΗ στη διαπραγματευτική ομάδα με μια εσωτερική προθεσμία για σχόλια που θέλετε να υποβληθούν στην Επιτροπή σε κάποια εποπτική αρχή. Βλέπετε εκεί πέρα το σχετικό φάκελο, τύπος ε, του μέτρου. Πατάτε εκεί πέρα και σας βγάζει το κάθε έγγραφο και το email με το οποίο βεβαίω σας στείλαμε όλα αυτά τα μέτρα. Και υπάρχουν όλες οι προθεσμίες λοιπόν. Τρίτον, κάποιες γενικές πληροφορίες ε, εκεί πέρα πάνω δεξιά. Συγκεκριμένα κατευθυντήριες γραμμές, ε, το τι κάνουμε με πράξεις κατεξιοδότηση και εφαρμοστικά μέτρα που έχουν εγκριθεί πρόσφατα από τους συντονιστές και δύο πίνακες ε, εποπτείας, ο ένας από την Γραμματεία και ο άλλος από την Κομισιόν για τις πράξεις που αναμένουμε ή έχουν ήδη φτάσει και τέλος δημιουργήσαμε φακέλους ε, με αρχεία τα βλέπετε στα δεξιά της σελίδας ε, ένας ε, φάκελος για κάθε οδηγία ή κανονισμό ο οποίος περιέχει κάποια εξουσιοδότηση. Πάρουμε ένα παράδειγμα. Αγορές και χρηματοπιστωτικά μέσα πατάτε στο φάκελο και βλέπετε τα σχετικά έγγραφα που έχει λάβει η γραμματεία και σας έχει στείλει από όταν ξεκινήσαμε αυτή τη σελίδα. Παραδείγματος χάρη διαβούλευση με, για την ΕΣΜΑ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πατάω πάνω στο έγγραφο και θα το δούμε. Αυτά βασικά. Ακόμα βεβαίως το δουλεύουμε, θα εξελιχθεί και άλλο. Θα λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σας και θα προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και αν έχετε κάποια ερώτηση ελάτε σε επαφή με την γραμματεία και θα σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το εργαλείο. Ελπίζω οι συνάδελφοι να το χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα για να δουλεύουμε πιο αποτελεσματικά και να γλιτώνουμε και χάρτη. Περνάμε τώρα στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι η ψηφοφορία για... με σύσταση να μην διατυπωθούν αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 εδάφιο 6 του κανονισμού με το οποίο το Κοινοβούλιο αποποιείται του δικαιώματο του να περάσουν τρεις ε, μήνες για να εξετάσει την πράξη αυτή. Αποφασίσαμε να προτείνουμε να μην ε, έχουμε αντιρρήσεις για μια πολύ συγκεκριμένη περιορισμένη πράξη ε, ε που αφορά το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και όχι το Ταμείο Εξυγίανσης, απλά αφορά το προσωρινό σύστημα προκαταβολών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών κατά τη διάρκεια της ε, προσωρινής περίοδου. Κάτι το οποίο πρέπει λοιπόν να ισχύσει το συντομότερο δυνατόν και νομίζω δεν είναι επίμαχο καθόλου. Η Κομισιόν για πρακτικούς λόγους μας ζήτησε να μην διατυπωθούν αντιρρήσεις και πρέπει να ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος. Μετά θα πάει στη διάσκεψη των Προέδρων, μετά από εκεί στην Ολομέλεια και αν το ζητήσουν 40 βουλευτές θα υπάρξει ψηφοφορία, αλλιώς θα πάει με την διαδικασία αυτή και θα τεθεί ενισχύ. Προετοιμάστε τις κάρτες σας γιατί η τελική ψηφοφορία θα είναι ηλεκτρονική. Θα ψηφίσουμε παραγράφους ε, εκτιμώντας ε, και αιτιολογικές σκέψεις. Οπότε μπορούμε νομίζω να τις ψηφίσουμε unblock, το πρώτο group και μετά πάμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμφωνείτε? Ωραία. Υπέρ. Αποχέ. αποχές εγκρίνεται τώρα να δοκιμάσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία δοκιμαστική δύο παραπάνω από τους σοσιαλιστές τρεις παραπάνω από τους σοσιαλιστές δύο τώρα παραπάνω ένας παραπάνω σας παρακαλώ κάποιος πρέπει να μην ψηφίσει. Ένας παραπάνω είναι ακόμα. Σοσιαλιστές. Μπορεί κάποιος να βγάλει την κάρτα του από σοσιαλιστές. Ωραία. Πέρας. Περνάμε τώρα στην κανονική ψηφοφορία. Τίθεται σε ψηφοφορία η απόφαση του να μην φέρουμε αντίρρηση στον κανονισμό της Κομισιόν της 8 Οκτωβρίου 2014 που αφορά το προσωρινό σύστημα προκαταβολών του ενιαίου Συμβουλίου Εξυγένσης. Και πέρας εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης το οποίο είναι πάρα πολύ σχετικό και σημαντικό ε, θέμα. Διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστοτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της τράπεζας. Μία πρόταση που είχαμε προτείνει πριν από το τέλος της προηγούμενης θητείας, αλλά το συζητάμε τώρα. Ο συγητής είναι ο κύριος Γκούναρ Χόκμαρκ και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω ορισμένες απόψεις για να δούμε πώς να προχωρήσουμε με αυτή την πράξη. Ευχαρίστως να συζητήσω περαιτέρω και με τους ε, κοινωνικούς εισηγητές και με όλα τα μέλη της Επιτροπής. Το σχέδιο είναι 18 Δεκεμβρίου να υποβληθεί το σχέδιο έκθεσης για να έχουμε ευχάριστα διάλειμμα για τα Χριστούγεννα. Τα σημεία αφετηρίας στα οποία θα βασιστώ θα ήθελα να τα μοιραστώ και μαζί σας. Πρώτα απ' όλα σήμερα είμαστε στο 2014 όχι το 2009 πλέον. Το 2009 ήταν ε, οξία η κρίση λόγω πολλών μακροοικονομικών ανισορροπιών αλλά και επειδή υπήρχε μια τεράστια έλλειψη απαραίτητων νομοθετικών πράξεων για να υπάρξει σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Νομίζω αυτό είναι σημαντικό να το διαπιστώσουμε ευθύ εξ αρχής διότι έκτοτε από το 2009 στο 2014 έχουμε κάνει πολλά. Βεβαίω, όπω και αν τοποθετηθεί κανεί, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, πολλά έχουν γίνει. Πολλοί κανονισμοί έχουν προβλεφθεί. Κάποιοι λένε ότι είναι υπερβολικά πολλοί, κάποιοι λένε το αντίθετο. Α μην όμω ε, παραμερίζουμε το γεγονό ότι οι κανονισμοί που προβλέφθηκαν είναι πολλοί το τοπίο του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην Ευρώπη έχει αλλάξει τελείως. Έχουμε και θα αναφέρω μόνο ακρόνημα και ας τα σκεφτείτε όλοι πώς θα τα ερμηνεύσετε. Έχουμε το ΕΜΙΡ, το ΜΙΦΙΝΤΙΟ, το CR, το CRD4, το DGS, το SRM, το SSM, όλα αυτά που γνωρίζετε. Έχουμε το EVR, όλες τις εποπτικές αρχές. Έχουμε μια εκβάθρον νέα διάρθρωση. Και είναι μια νέα διάρθρωση που δεν έχει ακόμα αρχίσει στην πραγματικότητα να λειτουργεί, γιατί είναι αρκετά πρόσφατη. Η εποπτεία, το νέο εγχειρίδιο κανόνων, το Single Rule Book, και μετά το SRM και το SSM, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγένσης και ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας. Και το BRD, δηλαδή η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγένση των τραπεζών. Δεν μπορώ να αποφύγω εδώ τα ακρόνημα. Ε, έχουν αλλάξει λοιπόν πολλά από την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε το 2009. Το άλλο που έχει αλλάξει είναι ότι έκτοτε από το 2009 η μεγαλύτερη μεταβολή στην ευρωπαϊκή οικονομία και έχει αυτό για μένα ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας είναι είτε το πιστεύετε είτε όχι οι αλλαγές στο έλλειμμα του προπολογισμού, ε, στο δημοσιονομικά ελλείμματα και η πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων. Εάν ε, σχηματίσει κανείς την καμπύλη σε ένα βάθος ε, ορίζοντα χρονικού, θα πούμε ότι έχουμε 900 δις ευρώ ε, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκρίνοντας με αυτό που λανσάρει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο κύριος Γιουνκέρ, 300 δηλαδή δις σε μια πενταετία. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά. Ε, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επενδύσει 900 δις ευρώ. Και αυτό πρέπει να το δούμε από την σκοπιά την εξή. Η υπόλοιπη, η υπόλοιπη παγκόσμια οικονομία μεγαλώνει, αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ασία. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε ότι αυτή η υποβάθμιση των επενδύσεων δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα να, ε, ως προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Εν τέλει μπορεί να μας οδηγήσει σε νέα οικονομική κρίση, διότι αν δεν επενδύσει κανείς εγκαίρος δεν θα διατηρήσει την ε, τα στοιχεία του ενεργητικού και την αξία τους που χρειάζονται για να διατηρηθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτά πάνε μαζί. Ξέρουμε λοιπόν ότι τα μεγάλα προβλήματα της οικονομικής κρίσης προκύπτουν όταν ακριβώς η αξία των στοιχείων του ενεργητικού πέφτει. Αυτό που φάνηκε για τα τεστ κόπωσης είναι ότι τα στοιχεία του ενεργητικού είναι ε, ιδιαίτερα σημαντικά. Αυτό είναι προφανές, αλλά πρέπει να το πούμε. Εάν οι αξίε αυτέ λοιπόν, οι τιμέ ε, συνεχώ μειώνονται, είναι πολύ δύσκολο να έχουμε απαιτήσει περκεφαλαίου, γιατί ακριβώ υπονομεύονται εξορισμού. Αυτά λοιπόν είναι δύο πολύ σημαντικά σημεία αφετηρία. Ένα τρίτο τώρα στοιχείο. Μια αντίδραση σε όλα αυτά. Η Ένωση των Αγορών Κεφαλαίων. Νομίζω αυτό είναι απαραίτητο, διότι η έλλειψη επενδύσεων είναι ουσιαστικά μια τάση που εμφανίζεται στι οικονομίε τη κρίση. Είναι προφανέ και αυτό. Ε, ισχύει για όλου μα. Ισχύει για τι οικονομίες ε, συνθήκε κρίση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε την απαραίτητη ρευστότητα για όλη την ευρωπαϊκή αγορά ώστε να έχουμε επενδύσεις και την ε, δημιουργία ρευστότητα ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό αυτήν την προοπτική βλέπουμε την διάρθρωση της νομοθεσίας για τις τράπεζες. Από αυτά τα τρία σημεία αφετηρίας. Θεωρώ άκρος σημαντικό να στηρίξουμε την έκφραση όλων αυτών σε μια ευρύθμως λειτουργούσα ε, ένωση των αγορών κεφαλαίων. Τι εννοούμε τώρα με την ένωση των αγορών κεφαλαίων. Πέραν του ενίου εγχειριδίου κανόνων θα μπορούσε να είναι ο μόνος ε, κατάλληλος φορέας ώστε να έχουμε ρευστότητα σε όλες τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω τα τεστ κόπωσης μας έδωσαν ακόμη περισσότερα στοιχεία περί αυτού. Οι κρίσει στις χρηματοπιστωτικές αγορές είχαν περισσότερο να κάνουν με την ε, λιανική και με τα μεσητικά, ε, με την αγορά κινήτων. Αυτό φάνηκε και από τα τεστ κόπωσης. Ε, φάνηκε ότι οι πολύ καταμένες τράπεζες είναι ούτως ή άλλως ένα πρόβλημα αυτές καθ' Αλλά μπορεί να δει κανείς τα πράγματα και αντιστρόφως. οι εξελίξεις στην Κύπρο θα είχαν αντιμετωπιστεί αλλιώς αν υπήρχαν τράπεζες εκτεταμένες. Εάν ε, εδώ το θέμα είναι ε, πώς θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά η πυραμίδα. Και έρχομαι τώρα στην οδηγία για την ε, ανάκαμψη και την εξυγίαση των τραπεζών οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν την ανθεκτικότητα και τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τα πλήγματα και όχι να ζητούν τα χρήματα των φορολογουμένων όταν τα προβλήματα προκύψουν. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτεταμένες τράπεζες που είναι και επενδυτικές και εμπορικές δεν, ε, δεν μπορεί να είναι αυτές καθεαυτές το πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν θέλουμε να είναι τα κριτήρια μας βασισμένα, βασισμένα στην διάρθρωση των τραπεζών ή στην ε, στον, παράγοντα του κινδύνου. Δηλαδή με το CRD4, το ΕΜΗ, το BRD ε, και όλη την υπόλοιπη νομοθεσία μας, οι συνολικές αυτές τράπεζες, οι εκτεταμένες αυτές τράπεζες τι δραστηριότητε τους, θα λειτουργούσαν διαφορετικά, αλλά θέλουμε να προκύψει και ασφάλεια από αυτή την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, διότι το ψυχολογικό κλίμα που δημιουργείται το γνωρίζουμε όλοι. Εάν μια τράπεζα βρεθεί σε δύσκολη θέση και το 8% που χρειάζεται για το bail αυτό θα επηρεάσει μόνο τους καταθέτες. Νομίζω είναι πολύ λίγες οι κυβερνήσεις που είναι σε θέση να ακολουθήσουν τις αρχές του κανονισμού για, που προκύπτουν ε, των κανόνων που προκύπτουν από την οδηγία BRD και το Μπέιλιν. Δεν νομίζω ότι ούτε στο Λονδίνο, ούτε στο Στοκχόλμη, ούτε στο Βερολίνο μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά. Οι κυβερνήσει δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα. Από αυτήν λοιπόν την προοπτική, νομίζω είναι σημαντικό να έχουμε ένα διαφοροποιημένο τραπεζικό σύστημα. αλλά ε, θέλουμε ένα τραπεζικό σύστημα που μπορεί να παράγει και ρευστότητα από την ε, λιανική πώληση υπηρεσιών στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Αλλά πρέπει να βασιστούμε στα κριτήρια ε, του παράγοντα κινδύνου. Νομίζω ότι οι συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, το proprietary trading, είναι κάτι σημαντικό που θα πρέπει να το ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή για την χρηματοοικονομική αγορά, την δημιουργία ρευστότητας. Πρέπει να έχουμε αυτή την προσέγγιση που είναι βασισμένη στον παράγοντα κινδύνου. Νομίζω στην νομοθεσία μας ε, με την BRD δίνουμε την ευκαιρία στις εθνικές αρχές να πούνε σε μια τράπεζα ότι δεν μπορείτε να εξηγενθείτε ούτε να διασωθείτε και πρέπει να αλλάξετε το επιχειρηματικό σας μοντέλο. Δηλαδή αυτό προκύπτει από το BRD. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε με αυτή την νομοθεσία ώστε να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε θα πρέπει ως σημείο αφετηρίας να αξιοποιήσουμε όλη την εποπτεία και όλη την νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι χρειαζόμαστε ένα εύρυθμο και ε, λειτουργικό ε, τραπεζικό σύστημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μας παρέχει ρευστότητα και χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Και θα πρέπει αυτό να διασυνδεθεί με την νομοθεσία που ήδη λειτουργεί, ώστε να έχουμε ένα σύστημα που μέσω του single rule book, του ενιαίου χειριδίου κανόνων, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη επενδύσεων και να επιστρέψουμε στην άνθηση των επενδύσεων και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Σιγητάλη, ο Πρόεδρος, για την εισήγησή σας. Πάρα πολύ σαφή οπότε θα είναι και ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και τώρα, ο Γιώργο Φρονβάης Τσέκερ, έχει το λόγο, ε, ο πρώτο εκ των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Κούναρ Χόκμαρκ για αυτήν την εντυπωσιακή του ε, εισαγωγή στο θέμα. Έχετε δίκιο 100% ότι χρειάζεται να δούμε το νομοθέτημα αυτό στα πλαίσια της νομοθεσίας που έχει προωθήσει τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή μας αλλά και άλλες επιτροπές. Και η πορεία αυτή της Γενικής Τράπεζας και αυτό που αποφάσισε δείχνουν γιατί μόνο για λίγες τράπεζες χρειάζονται παραπάνω χρήματα και δεν είναι κάτι θέμα μεγάλης κλίμακος. Όλα αυτά που έγιναν όταν ολοκληρώθηκαν τα stress test Οπότε βλέπουμε αν θα χρονίσει όχι αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε και αλλού στον κόσμο ότι τώρα επεξεργάζονται πιο δυναμικές λύσεις από την Eurozone και όχι υπάρχει ανάπτυξη πιο γρήγορη. Οπότε βλέπουμε γιατί τώρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα. Υπάρχει τώρα ένα συγκεκριμένο μέτρο θέλω να σε την προσοχή. Είναι αυτού του είδους η χαμηλό ρυθμού μόχλευση. Η οποία όμως να είναι συνεχούς μορφής. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πολύ όταν φτάσουν τα πράγματα στο χειρότερο. Αν έχουμε λοιπόν κάτω από 3% μόχλευση, τότε κανείς ξαναπέφτει σε κατάσταση κρίσης σαν τράπεζα. Οπότε βλέπουμε αυτά τα λάθη τα οποία για κάποιο τρόπο είναι υγιεινή στο σημερινό σύστημα και που πάνε να τρυπώσουν και στην μεταρρύθμιση αυτή. Ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Θέλουμε να είναι πιο ανθεκτικό το σύστημα το τραπεζικό. Έναντι των κινδύνων για κάποιες αποφάσεις που οι εποπτικές αρχές και οι κυβερνήσεις όπως είπατε ε, βρίσκονται υποπίεση να λάβουν για να προβούν σε ακόμα μια διάσωση, άρα το σύστημα να γίνει πιο ανθεκτικό. Και σε αυτά τα πλαίσια Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία. Δεν είμαι καν βέβαιος ότι κάνουμε αρκετά με αυτά που κάνουμε. Να σας πω δύο παραδείγματα όπου θα σας δείξω τι εννοώ πρώτα πρώτα την απαγόρευση κάποιων δραστηριοτήτων. Αν μια ματιά ε, στην πρόταση νόμου ιδίω όσον αφορά την απαγόρευση του proprietary trading των συναλλαγών ιδίου λογαριασμού Βλέπετε γιατί χρειάζεται αυτή η μόχλευση που μπορούν δηλαδή οι τράπεζες αυτή την περίπτωση να δανείσουν. Και αυτό δεν ήταν η τελευταία, δεν έγινε η τελευταία κρίση, αλλά είναι μια κρίση που σου και πάρα πολύ καιρό για τις τράπεζες. Να λοιπόν γιατί ξαφνικά δεν μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας εύκολα αλλά από την άλλη μεριά και εγώ δεν βρουν μια λύση γιατί πάρα πολλέ μεγάλε τράπεζε όπω το Citigroup δανείζουν σε capital management αλλά βρέθηκαν τελικά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τώρα. Να, που οδήγησε η απαγόρευση. Δεν είναι τόσο σημαντικό για την ε, πραγματική οικονομία το αν ε, θα επιτρέψουν στι τράπεζε να κάνουν αυτά τα, να δίνουν αυτά τα δάνεια τέλο πάντων. Βλέπουμε μόνο τι θα μπορούσε να διορθωθεί σε αυτό το νομοθέτημα τώρα και κάτι άλλο τώρα. Αν και έχω πολλά που θα μπορούσα να πω είναι το θέμα της διακριτικής ευχέρειας. Ναι αυτή τη νομοθεσία που έχουμε τώρα, έχουμε πολλά επίπεδα, ούτε μπορούμε να δούμε τι κριτήρια χρησιμοποιεί η, ε, ο φορέας αυτός για τις τράπεζες και τελικά είναι στη κρατική ευχέρεια της Ευρωπαϊκής Αρχής να λάβει κάποιες αποφάσεις επί τη βάση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από κάποιους άλλους εμπλεγωμένους. Και εκ των υστέρων γίνεται η διαπίστωση του κατά πόσον αυτό είναι επαρκές. Και βλέπουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ένωση Τραπεζών, η Υποπτική Αρχή, όλοι αυτοί οι τρεις ε, είναι καλόπιστοι γιατί στριμώχονται πάρα πολύ ακριβώς λόγω των πιέσεων από τους λομπίστες. Μα και εμείς πιεζόμαστε από τα λόμπι στην Επιτροπή μας. Άρα θα πρέπει να βοηθήσουμε λιγάκι με κάποιες διαδικασίες που να μπορούν να αποτελούν κάτι σαν δίχτυα ασφαλείας ότι ναι, καλά τα πάρει, χρειάζονται όλα αυτά που κάνετε, αλλά να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή ούτως πίν, που κανείς δεν θα μπορεί να την ε, περάσει. Και δεν μιλάμε για οποιαδήποτε τράπεζα, μιλάμε για τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης. Άρα θα υπάρχει αυτό το όριο. Θα λέμε ότι μέχρι εκεί μπορείτε να πάτε και όχι παραπέρα. όλα αυτά. Και μπορούσα να πω και πολλά άλλα, δεν έχω το χρόνο. Πρόκειται απλώ για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Να σας δώσω έτσι μια πρόγευση του πού θα πάμε αυτή την νομοθεσία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος τώρα, ο μιλητής για την ECR είναι ο Σαΐτ Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω αυτό το είχαμε συζητήσει κύριε. την τελευταία θητεία οι πολιτικέ ομάδε όμως ότι ας και ας μην συμφωνούμε πρέπει κάτι να κάνουμε. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε κάποιος κοινό παρονομαστής σε αυτή την τελευταία θητεία όπου είχαμε την έκθεση Μακάρθη και ω επιτοπλίστων συμφώνησαν όλο, το πολιτικό φάσμα του Κοινοβουλίου. Όπως είπε και ο Γκούνα, να δούμε τι γίνεται με τι εποπτικές αρχές, τι γίνεται με όλα αυτά τα αρχικά λύσαν το πρόβλημα. Ούτως ώστε να σωθούν οι τράπεζες που αυτό κοστίζει χρήματα στους φορολογουμένους. Άρα θα πρέπει κάτι να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα και να μην γλιστράμε σε ε, λαϊκιστικές θέσεις, να, ε, να ε, επιτιθέμεθα στα hedge funds γιατί τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Κάποιες χώρες μπόρεσαν να σωθούν από τη χρεοκοπία, αλλά κάποιες τράπεζες όχι. Κάπως τώρα θα βάζω όλα στο ίδιο σακί, αλλά δεν έχουμε τώρα το χρόνο να εξειδικεύσουμε. Έχουμε επομένω κάποιε προτάσει που επιφωνησαν πολλε πολλέ πολιτικέ ομάδε. Πρώτα-πρώτα είπαμε ότι αν κάποια ε, τράπεζα πτωχεύσει, τότε α την αφήσουμε στην τύχη τη και όχι να ε, κάνουμε τον κόσμο να τη σώσει. Να τη θα πει ε, σε μια ελεύθερη αγορά, οικονομική επιστήμη. Γιατί ο φορολογούμενος να σώζει μια τράπεζα. Την αφήνουμε να πτωχεύσει. Αυτό θα πει αγορά με ανταγωνισμό. Γιατί οι φορολογούμενοι είναι να το κάνω αυτό. Θα πρέπει τα χρήματα των φορολογουμένων να διατίθενται σε άλλους σκοπούς. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε είναι το θέμα της ευθύνης. Συμφωνώ όπως και αριστερά ότι θα βρήκαμε να τα χρήματα όταν όλα πάνε καλά, αλλά όμω το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Τώρα κάτι άλλο και ελπίζω ότι σε αυτή τη θητεία θα το συζητήσουμε είναι το τι γίνεται ναι, την λογοδοσία ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για... στον ισολογισμό, δεν υπάρχει πρόβλεψη για μεγάλες ζημίες και όταν έχουμε κάποια έκθεση προβολή των τραπεζών με τα CDS και με άλλους τρόπους γιατί σήμερα η λογιστική του το επιτρέπει αυτό στις τράπεζες. Άρα θα πρέπει να δούμε μέχρι πού μπορεί να γίνει αυτό, να ισχύσει αυτό και αυτό θα πρέπει να το κρίνουμε στην Επιτροπή μας. Αυτό θα πρέπει να λύσουμε σαν πρόβλημα. Οπότε όταν κάποια τράπεζα να δούμε όλα αυτά τα, τα αρχικά έχουν βοηθήσει, μπορούν να βοηθήσουν. Θα πρέπει να έχουμε οποιαδήποτε ε, συμβολή του φορολογουμένου. Τι είδους παρέμβαση θα πρέπει να γίνεται. Ιδανικό για μένα θα ήταν το ότι όποια τράπεζα είναι να πτωχεύσει, ας πτωχεύσει. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εκαθάρισης, ε, σύνδυγη κλπ και έτσι να μπορούν οι καταθέτες να πάρουν τα χρήματά τους ε, για να ζήσουν προς τους λογαριασμούς τους, αλλιώς πάμε σε κοινωνική αναταραχή. Επίσης, τι γίνεται με τις παγκόσμιες τράπεζες, να ωφελούνται από κάποιες ενισχύσεις και επιδοτήσεις. Ξέρω ότι θέλει παγκόσμιες τράπεζες ο Γκούναρ, αλλά τελικά με αυτά τα χρήματα της διάσωσης ποιον βοηθάμε. Βοηθάμε κάποια δραστηριότητα μήπως που δεν θα έπρεπε να τη βοηθούμε γιατί πρόκειται για χρήματα φορολογούμενα. Άλλο. Να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο από ό,τι θέλουμε να θεσμοθετήσουμε να μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω, να μην σταματάμε αυτά τα κράτη. Όποιος θέλει να προχωρήσει μόνος, μα προχωρήσει γιατί σε κάποια κρατημέλη κάποιες μεταρρυθμίσεις συζητούνται και υπάρχουν επομένως κάποιες προτάσεις από αυτά τα κρατημέλη. Οπότε να συνεργαστούμε με συναδέλφους που έχουν ασχοληθεί την τελευταία θητεία με το ίδιο θέμα. Οπότε, τη συνένεση που τότε είχαμε διαμορφώσει, ας την συνεχίσουμε και σε αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ. Thank you. Now for the ALDE group. Ευχαριστώ. Σιλβί Γκουλάρ για την άλλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα περιμένω να βάλουν όλοι τα ακουστικά τους. Ωραία. Είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και κατά την άποψή μου είναι πιο σημαντικό ακόμη να είμαστε συνετοί τώρα επειδή υπάρχει και μια νέα επιτροπή που ανέλαβε. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο νέος επίτροπος θα προθέσει το όλο κείμενο ως δι. Επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν αντιστάσεις από το Συμβούλιο και οι εμπειρίες που είχα από τον τριμερή διάλογο μου έχουν δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο εάν έχουμε τέσσερις στήλε στον ε, τριμερή διάλογο, ε, να ακολουθήσω τη συλλογιστική του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο. Και κυρίως θα ήθελα και την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αυτό το ε, κείμενο. Διότι όλη η συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εποπτείας πολύ σημαντικές αρμοδιότητες. Υπάρχει ε, σήμερα αρχίζει και αναλαμβάνει καθήκοντα το SSM. Θα δούμε τι θα κάνει από εδώ και στο εξή. Είδαμε μάλιστα μια πρώτη, ένα πρώτο δείγμα από τα τεστ κοπόσεω, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να τα θέσουμε όλα σε μια αρχή που μπορεί να μα πει κάποια στιγμή ότι δεν έχετε τη δυνατότητα ή ε, τη διάθεση να τα φέρει ει πέρα. Τώρα, ω προ το Ταμείο. Ε, Έχουμε τρία στοιχεία, αλλά θα πρέπει έτσι κι ε, σε αυτό το χρονικό σημείο να τα συζητήσουμε περαιτέρω και θα τα δούμε και με τον εισηγητή και με του κοιόδη. Το πρώτο σημείο λοιπόν ανησυχία είναι ο κατακαιρματισμό τη ε, εσωτερική αγορά. Στο κείμενο αυτό ε, αναφέρεται η ιδέα βάσει του Ταμείου να ισχύει η νομοθεσία των κρατών μελών και όχι μια κοινή. Εκεί μπορεί να υπάρχουν αποκλήσει. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν προβλέψει όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, Γερμανία ή το υπάρχουν προβλέψεις για το θέμα αυτό, αλλά αυτό δεν είναι αυτό καθε αυτό πρόβλημα εάν καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα και δεν καταστρέφουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των ε, διαφόρων κρατών ή των τραπεζών όπου έχουν την έδρα τους εκεί. Αυτό ε, δεν θα διευκολύνει απαραίτητο και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ε, με ένα single rule book που μπορεί να γίνει μέρο τη εθνική νομοθεσία. Αλλά τέλο πάντων αυτό θα το δούμε. Θα δούμε πώ θα νομοθετήσουμε. Έχουμε ήδη ζήσει με το σχετικό κανονισμό και είδαμε με αυτή την αφορμή ότι υπήρχε ένα τεράστιο πειρασμός εθνικοποίησης ε, είτε των κανόνων είτε των κονδυλίων. Να προσέξουμε λοιπόν πάρα πολύ εδώ την ενότητα της εσωτερικής αγοράς έχοντας υπόψη και ένα άλλο στοιχείο που πολλές φορές ε, <coughs> επηρεάζει την δική μας νομοθεσία. Ένα πρόβλημα δημοκρατικό, ε, βαθύ δημοκρατικό μάλιστα πρόβλημα και χαίρομαι που μπορώ να το σημειώσω εδώ, δηλαδή από πού προέρχονται τα κείμενα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Βλέπουμε το CDR4 το ξαναβλέπει με το ΤΙΛΑΚ, το ε, Συμβούλιο Δημοσιονομική Σταθερότητα και βλέπουμε να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων εθνικών ή διεθνών και δεν ξέρουμε όλα αυτά πώ συνδυάζονται μεταξύ του. Δεύτερο σημείο ανησυχία, το ανέφερε ο συνάδελφο και είναι αρκετά προφανέ, πώ θα καταπολεμήσουμε τον υπερβολικό κίνδυνο πώς μπορούμε ε, να αποφύγουμε την στήριξη από τους φορολογουμένους λόγου χάρη. Ακόμη και αν λέει ο κύριος Κέλλαμ αυτό που είπε, είναι τράπεζες στον ΕΒ που έχουν εθνικοποιηθεί πάνω από 80%. Ας ε, αποφύγουμε λοιπόν αυτήν την ε, κούρσα προς το χρήμα των φορολογουμένων. Βλέπουμε ότι στις αντικές κρίσεις έχουν την αντίθετη τάση τα κρατημέλη. Δηλαδή όταν οι υπουργοί οικονομικών να βρίσκονται σε δύσκολη θέση σκέφτονται να σώσουν πρώτα τις τράπεζες. Ακόμη και όταν το κόστος είναι μεγάλο, ακόμη και όταν είναι ε, αμύθιτο το ποσό. Ας μην είμαστε λοιπόν εδώ αφελείς. Πρέπει να γίνει μια αλλαγή πολύ ριζοσπαστική όπως έγινε με το SRM και το SSM. Ε, ε, και εδώ περιμένω να δω τι θα γίνει όταν μια μεγάλη τράπεζα έχει σοβαρό πρόβλημα και κλονίζεται. Δεν, και κλειδονίζεται μάλλον. Δεν ξέρω, ε, δεν, δεν λέω να μην τα σκεφτούμε καθόλου αυτά, απλώς να σκεφτούμε τι ε, πολύ έντονες, τις ε, κραυγαλαίες αντιστάσεις που υπάρχουν στο Συμβούλιο των Υπουργών εδώ ω προ αυτά. Και... Ε, Ποια θα είναι η ισορροπία μεταξύ του υπερβολικού κινδύνου και την προάσπιση της άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων από τις ε, τράπεζες. Είδαμε ότι ε, στις γραπτές απαντήσεις του υπευθύνου που ήρθε να μας μιλήσει, ε, είδαμε τι έχει στο μυαλό του οι δραστηριότητε κάποιων τραπεζών τη Ευρωζώνη που ήδη κάνουν, δίνουν μεγαλύτερη στήριξη σε μεγάλε επιχειρήσει ή μικρομεσαίε που εκδίδουν ομόλογα. Εδώ Πώς θα τα καλύψουμε αυτά τη στιγμή που έχουμε απελπιστική ανάγκη επενδύσεων και ανάπτυξης. Πώς θα εμποδίσουμε να γίνουν αυτά με ιδίως ως ρόλο των τραπεζών. Και αν δεν το κάνουν οι τράπεζες, πώς θα αποφύγουμε να περάσουμε στο παράλληλο τραπεζικό σύστημα, στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Ε, εδώ θα τα παρακολουθούμε στενά όλα αυτά, διότι δεν είναι καθόλου προφανές να βρούμε τους κατάλληλους ορισμούς του τι απαγορεύεται και τι όχι. Και η τελευταία μου, το τελευταίο σημείο ανησυχία, θα έλεγα ότι είναι κάπω ακαδημαϊκή και φιλοσοφική ανησυχία μου. Δηλαδή, θα ήθελα να βρεθούμε σε μια ε, κατάσταση που τη γνωρίζει πολύ καλά η ανθρωπότητα, να προσπαθούμε να διαχωρίσουμε το καλό από το κακό. Ο πειρασμό είναι να υπάρχει αυτό ο απόλυτο μανιχαϊσμό. Δηλαδή, κάποιοι να λένε ότι υπάρχουν κακέ τραπεζικέ δραστηριότητε θα πρέπει να τι διαχωρίσουμε από τι καλέ τις ενάρετες ε, τραπεζικές δραστηριότητες. Αυτή είναι μια τάση της ανθρώπινης φύσης που δεν μας έχει πάει και πολύ μακριά. Εγώ ξέρω και πιο καλό πολιτικό που μου είχε πει «Σκασίλα μου μεγάλη, αρκεί να πούμε ότι κάτι καταφέραμε». Νομίζω ότι αυτή τη θεώρηση που από φιλοσοφική άποψη μπορεί να είναι κάπω αμφίβολη, ε, ελπίζω ότι μοιράζονται πολλοί συναδελφοί εδώ, αλλά τουλάχιστον να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που να είναι κάπω ε, ε, θετικό μάλλον. Ε, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό λοιπόν τη ενιαία αγορά, να δούμε πώ από οικονομικέ απόψει θα καλύψουμε τον υπερπολικό κίνδυνο και επίση να προστατεύσουμε και τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματο, χωρί να έχουμε την ψευδέστηση ότι διαχωρίσουμε το καλό από το κακό. και ότι θα διευθετήσουμε πλήρω το όλο πρόβλημα. Τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα στην πραγματικότητα και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι όχι απλώ μα περιμένουν οι ακροάσει ε, που θα ακολουθήσουν. Πρέπει να, να ακούσουμε και τον κύριο Λικάνεν, ε, ο οποίο ξέρουμε ότι θα επηρεάσει αυτά τα πράγματα, αλλά και όλου του υπευθύνου του κλάδου που θα καθορίσουν την πορεία των πραγμάτων. Και να πω για τι μεγάλε αυτέ τράπεζε, τι παγκόσμιες ιδιαίτερα τι μεικτέ τράπεζε, δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να απαγορεύσουμε ένα τραπεζικό μοντέλο, απλώς κάποιες πρακτικές ίσως να πρέπει να αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Γκουε Φάμπιο Ντεμάσιμο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Χέκμαρκ για την έκθεσή σας. Πρώτα απ' όλα να σας ε, πω κάτι το οποίο ίσως φανεί περίεργο. Ε, ως αριστερός εμένα μου αρέσουν τράπεζες, αλλά οι βαρετές τράπεζες. Παλιά είχαμε τον λεγόμενο κανόνα 3-5-3. Δηλαδή ο τραπεζίτης ε, δάνιζε με, δανειζόταν με 3%, δάνιζε με 5% και στις 3 η ώρα σχολούσε και πήγαινε για γκολφ. Σήμερα λοιπόν το βασικό πρόβλημα του κυρίου Χόκμαρτ. Ο κ. Κόκκινοφ μα λέει πω ε, το βασικό πρόβλημα το οποίο προκαλεί την έλλειψη πίστης για τι επενδύσει είναι οι υπερβολικέ ε, ρυθμίσει. Πράγματι έχουμε όλε αυτέ τις ρυθμίσει που λέτε, μύφητη και τα λοιπά, αλλά σημασία δεν έχει ο αριθμό ε, των ρυθμίσεων, αλλά το είδο του. Και θέλω εγώ να πω πω η νομοθεσία είχε 37 σελίδε. ο νόμος Dodd-Frank είχε 800 και δεν ξέρω πόσε σελίδε έχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά σημασία έχει να είναι πραγματικά αξιόπιστη. Και εδώ πέρα πραγματικά έχουμε φτάσει στην στιγμή της αλήθειας. Ε, εδώ πέρα θα κρυθεί όλη μας η νομοθεσία. Το ανέφεραν ήδη οι συναδελφοί μου. Έχουμε το πρόβλημα των εταιριών που είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν, οπότε ε, οτιδήποτε και αν αποφασίσουμε για τη συμμετοχή των καταστών δεν θα υπάρξει τέτοια πράγμα σε τράπεζες που είναι πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν γιατί ακριβώς κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και υπάρχει ήδη εξαίρεση αυτή ήδη σήμερα στην νομοθεσία. Οπότε αυτή η υπόσχεση είναι μια υπόσχεση η οποία δεν ισχύει, ότι δηλαδή δεν θα ξαναπληρώσει ποτέ ο φορολογούμενος για ε, τράπεζες που είναι πάρα πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν. Επίσης διαφωνώ, εάν το πρόβλημα ήταν οι υπερβολικές ρυθμίσεις, αν δούμε την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου δεν υπάρχει αρκετή πίστοση για πραγματικές επενδύσεις από τις τράπεζες, ο λόγος θα ήταν πως οι ελληνικές και οι ιταλικές τράπεζες αντιμετωπίζουν υπερβολική ρυθμίση. Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οπωσδήποτε υπάρχει πάρα πολύ σημαντική σχέση ε, μεταξύ της μακροοικονομίας και των τραπεζών. Δεν μπορούμε να έχουμε υγιή οικονομία χωρίς υγιείς τράπεζες, αλλά και αντιστρόφως. Τότε, αν δεν, υπάρχουν αρκετέ, αν δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση για επενδύσεις, δεν θα υπάρχει και ε, πίστοση από τις τράπεζες. Τρίτον, ε, Μιλάμε πάρα πολύ για παράγωγα, δημιουργία αγορών κτλ. Και οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους χρειάζεται αυτό. Αλλά αν δείτε τα στοιχεία δεν μπορούμε, αν δείτε τα στοιχεία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το τι γίνεται στα παράγωγα μόνο από την πλευρά του hedging, δημιουργίας αγορών κτλ. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Υπάρχει τόσο μεγάλη αύξηση πλέον ε, των ε, της ε, πλευράς ε, του trading των τραπεζών και με τα παράγωγα βεβαίω δεν απομονώνεται κανείς από τον κίνδυνο. Οπότε, οι πρώτες μου σκέψεις εδώ πέρα πηγαίνουν προς την κατεύθυνση του Τζέικομπ. Πρέπει να μιλήσουμε για τον ε, σκιώδη τραπεζικό τομέα, δανεισμό σε hedge funds το επίπεδο επίσης ε, διακριτικής ευχέρειας ε, που υπάρχει. Δεν θέλουμε να υπάρχει lobbying ε, και πολιτική πίεση στις εποπτικές αρχές, οπότε πρέπει να είναι σαφείς οι κανόνες, λιγότερη διακριτική ευχέρεια, είτε μιλάμε για το μέγεθος των χαρτοφυλακίων ή άλλα μέτρα και βεβαίως πρέπει να φύγουμε από αυτά τα εσωτερικά μοντέλα ε, που βασίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου. Γιατί και πριν βασιζόμασταν όντως στα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών που έχουν που απέτυχαν τόσο εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης και πραγματικά δεν λύσαμε εδώ πέρα το πρόβλημα στην ουσία του. Τελευταίο σχόλιο Υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι στο νομοθέτημα αυτό, στο πρώτο άρθρο, καλοί στόχοι και θεωρούμε πως το θέμα του διαχωρισμού πρέπει να αφορά όλους αυτούς τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και όχι μόνο στον αυτόν τον γενικό και αόριστο ορισμό της απειλής ε, της ε, σταθερότητας. Και άρα στο πλαίσιο αυτό θα παρατηρήσουμε την πρόοδο της σχετικής νομοθεσίας και τώρα πρέπει πραγματικά να επιδείξουμε αποτελέσματα στους φορολογούμενους και εμείς θα φροντίσουμε να μην αθετήσουμε αυτή την υπόσχεση. Σας ευχαριστώ. Για τους πράσινους Φίλιπ Λάμπερτς. Ναι Φάμπιο είμαι σίγουρος πως θα κάνετε περισσότερα από το να παρακολουθήσετε τις εξελίξεις και συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είπε ο Γιάκοβ και από αυτά που είπε ο Φάμπιο και η Σιλβή και ο Γκούνερ. Να ξεκινήσω λέγοντας πως ε, συμφωνώ με κάτι το οποίο είπε ο Γκούνερ, η Ευρώπη υποφέρει από μεγάλη έλλειψη επενδύσεων, ε, δηλαδή χρήματα τα οποία θα επενδύονται μακροπρόθεσμα με υπομονή και από τον ιδιωτικό και από τον δημόσιο τομέα. Ε, ακούμε τώρα πως οι πολλές ε, ρυθμίσεις βλάπτουν τις ε, επενδύσεις. Εντάξει, μπορεί να μην είναι μαγική λύση η μεταρρύθμιση του τομέα, αλλά οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Αν δούμε παραδείγματο χάρη την νομοθεσία Glass-Steagall, εάν μαζεύει κανείς ε, καταθέσεις δεν έχει να τις κάνει τίποτα άλλο παρά να τις επενδύσει στην πραγματική οικονομία. Ούτε δραχμή από αυτά τα οποία μαζεύει δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Άρα, εάν υποθέσουμε πως μέρος των καταθέσεων πηγαίνει για άλλες χρήσεις, τότε χωρίς ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, πράγματι εμποδίζουμε τις επενδύσεις γιατί μειώνουμε το χρήμα το οποίο πηγαίνει στην πραγματική οικονομία. Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνείς, Σιλβία, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων, Glass-Steagall δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς τώρα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, οι τράπεζες που ήταν και επενδυτικές και λιανικές ε, δεν ήταν το πρόβλημα. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και εγώ θέλω λίγο να... Και θέλω πράγματι να έχουμε ε, ένα ε, σύστημα το οποίο θα έχει ποικιλομορφία. Υπάρχει η θέση για τράπεζες που θα κάνουν τα πάντα. Αλλά πόσο μεγάλες πρέπει να είναι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Η δέξια ε, και η φορτής στη χώρα μου. Εάν υπήρχε ένας δομικός διαχωρισμός, η φορτής δεν θα είχε 45 δισεκατομμύρια άχρηστα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό τους. Γιατί μου λέτε πως ε, οι τράπεζες που τα κάνουν όλα έχουν πρόβλημα και η Goldman Sachs ε, ε, ήταν μόνο επενδυτική τράπεζα και τα κάχα στην Ισπανία ήταν μόνο τράπεζες λιανικής. Ναι, αυτά ισχύουν, αλλά η απάντηση είναι οι τράπεζες που τα κάνουν όλα. Εδώ πέρα δηλαδή διαφωνεί η πραγματικότητα. Τέταρτον, έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά. Υπάρχει υπερβολικά πολυνομοθεσία και εδώ πέρα συμφωνώ με τον Σαΐδ. Κοιτάξτε, εγώ τα μετράω τα πράγματα με έναν απλό τρόπο και έχω μια φιλελεύθερη προσέγγιση ως προς αυτό. Ζούμε σε μια οικονομία τη αγορά. και δεν μπορώ να συμφωνήσω πως οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία να έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς και τι κάνει, κορώνα κερδίζει, γράμματα χάνουν οι άλλοι. Αυτό δεν είναι η οικονομία της αγοράς, είναι η σοβιετική οικονομία. Και κατά την άποψή μου θα τελειώσουμε με όλες αυτές τις ρυθμίσεις όταν μπορούμε πραγματικά να κοιτάξουμε στα μάτια τους φορολογούμενους και να τους πούμε πως δεν υπάρχουν πλέον ε, τραπεζικά ιδρύματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα για να χρεοκοπήσουν. Και πράγματι η οδηγία Κεφαλαιακών απαιτήσεων κάτι βάζει ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση και λίγο παραπέρα. Αλλά απέχουμε ακόμα πολύ. Και πάλι πρέπει να αποφασίσουμε με ποια πλευρά είμαστε. Είμαστε υπέρ μιας οικονομίας αγοράς ή όχι. Αλλά δεν μπορούμε να θέμε η οικονομία της αγοράς όταν μας συμφέρει και μετά ρυθμιστική και κρατικιστική οικονομία όταν δεν μας συμφέρει ή το ένα ή το άλλο, έτσι. Αυτές ε, ήταν οι πρώτες μου παρατηρήσεις. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποια άρθρα ε, στα οποία θεωρούν πως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Πρώτα απ' όλα για τους στόχους της νομοθεσίας. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε και απευθύνομαι εδώ πέρα στη Σιλβή. Δεν είναι οι κακές οι τράπεζες λιανικής και οι καλές τράπεζες λιανικής και οι κακές επενδυτικές τράπεζες. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και τράπεζες λιανικής που έχουν κάκιστη διαχείριση. Αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε είναι την μετάδοση όταν έχουμε πρόβλημα σε ένα τμήμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος να μην μεταδίδεται αλλού. Και δεύτερον, δεν θέλουμε επιδοτήσεις του κράτους σε πράγματα τα οποία δεν είναι οι βασικές τραπεζικές λειτουργίες που είναι ουσιαστικές για τη λειτουργία της κοινωνίας. Δηλαδή υπάρχει μια δημόσια εγγύηση για τις βασικές δραστηριότητες ε, άμα το κάνουμε αυτό δηλαδή εγώ θα έλεγα να τις κάνει και το κράτος αλλά τέλος πάντων να περιορίσουμε τις επιδοτήσεις σε δραστηριότητες που είναι ε, ουσιαστικές για την οικονομία και εκεί πέρα πρέπει να είμαστε σαφείς στον ορισμό των δραστηριοτήτων αυτών που θεωρούνται πραγματικά ε, κέρια σημασία και των λοιπόν. Και πραγματικά, αν θέλουν να παίξουν οι μέτοχοι των τραπεζών, να το κάνουν, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά με την ε, δικιά τους την τσέπη. Έτσι, και δεν είναι δυνατόν με τα λεφτά των δημοσίων επιδοτήσεων να κάνουν αυτά τα οποία θέλουν. Δεύτερον, στο άρθρο 3, το πεδίο εφαρμογή. Η πρόταση ισχύει για περίπου 30 τράπεζες. Εμείς θεωρούμε πως πρέπει να πάρουμε τον ορισμό που υπήρχε στην Τραπεζική Ένωση για το, που λέει τι, ποια τράπεζα είναι σημαντική και να την εφαρμόσουμε και στα 28 κράτη-μέλη. Οπότε, 134 ε, της Ευρωζώνης συν ε, εκτός της Ευρωζώνης όσες εμπίπτουν σε αυτόν τον ορισμό για να έχουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό γιατί μπορεί να λέτε ναι κάποιες από αυτές τις τράπεζες ε, δεν ε, δραστηριοποιούνται στις χρηματαγορές, ναι αλλά τα πράγματα αλλάζουν, έτσι δεν είναι στατική η κατάσταση, είναι δυναμική και θέλουμε να μην ε, μπουν σε επικίνδυνα νερά οι φυστάμενες τράπεζες. Για το για ίδιον εγώ θεωρώ πως πρέπει να τα απαγορεύσουμε, αλλά εν περιπτώσει τώρα. Το πώς θα το διακρίνουμε από οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή είναι τι, να βάλουμε ένα τσιπάκι στον εγκέφαλο κάθε trader για να δούμε τι κίνητρο έχει. Δεν είμαι υπέρ, μάλλον παραβιάζουμε εδώ πέρα κάποια δικαιώματα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε έχω έναν αρκετά ευρύ ορισμό για το τι είναι συναλλαγή ε, για ίδιον Οπότε μετά διαχωρισμός άρθρο 2.21 συμφωνούμε με τα βασικά στοιχεία αλλά αυτό το οποίο θα προτιμούσαμε είναι αν θέλετε ένα σύστημα με κάποιες βαθμίδες. Δηλαδή κόκκινο θα είναι υποχρεωτικός διαχωρισμός, πράσινο προφανώς εάν είσαι κάτω από αυτό το κατόφλι πάλι δεν το συζητάμε καν και μετά το κίτρινο που παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, πιθανότερα υψηλότερος λόγος κεφαλαίου και κάποια διακριτική ευχέρεια, αλλά όπως είπε ο Φάμπιο, η διακριτική ευχέρεια εντός πλαισίων. Δεν θέλουμε οι τράπεζες να διαπραγματεύονται ε, και να κάνουν συναλλαγές για διονόφιλος με τις ε, επιδοτήσεις ε κατά κανόνα. Εάν δούμε ε, το πώς θα μετρήσουμε παραδείγματο χάρη το κόστος το οποίο χρησιμοποιείται για συναλλαγές ε, με το ρίσκο αντισυμβαλωμένου, τι να πω τώρα για το βασικό κύριο ίδιο κεφάλαιο θα έλεγα πως είναι ένα 10%, τα, το κύριο ίδιο κεφάλαιο 5%, Έχουμε πάρα πολλέ επιφυλάξεις σε μπάση περιπτώσει. Ξέρω πως τα stress test ε, αυτό χρησιμοποιούσαν ω μέτρο το οποίο είναι τελείω λάθος. Έχω δει άλλε μελέτες που από τα ίδια δεδομένα βγάζουν ε, άλλα συμπεράσματα, λένε πως χρειάζεται πολύ περισσότερο κεφάλαιο για να επιβιώσουν οι τράπεζες. Και τέλος, εδώ πέρα συμφωνώ με την ανησυχία της ε, Σιλβή, έχουμε τις εξαιρέσεις για τα κράτη-μέλη. Κοιτάξτε, αν μία χώρα τα έχει πάρει σοβαρά αυτά, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ ας πω συχνά κριτική, αλλά εδώ πέρα μάλλον φτάνουν με τη μεταρρύθμιση Vickers πάρα πολύ κοντά στο χρυσό κανόνα. Η άποψή μου για τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη Γερμανία, στο Βέλγιο και στη Γαλλία, τι ήταν αυτά κατά βάση ελιγμοί που δεν επέτυχαν κανένα διαχωρισμό, αλλά είχαν στόχο να προλάβουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σου Σιλβί πως πρέπει να διαφυλάξουμε την ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια επιλογή που πρέπει να γίνει και είναι δύσκολη. Είτε το τίμημα της ενιαίας αγοράς είναι να κάνουμε ψευδείς μεταρρυθμίσεις όπως στη Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ ως τίμημα ή και βεβαίως μετά πρέπει να διατηρήσουμε την εξαίρεση των Βρετανών για να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν ή φέρνουμε το επίπεδο των Βρετανών στην Ευρώπη και μετά διατηρούμε την ενιαία αγορά. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Αλλά δεν είμαι διατεθειμένος εγώ να θυσιάσω τον στόχο της μεταρρύθμισης για την ενιαία αγορά. Δηλαδή μια στραβή, στρεβλή ενιαία αγορά δεν είναι καλύτερη από μια ενιαία αγορά όπου τουλάχιστον ε, ένα νησί προσπαθεί να διατηρήσει την οικονομία της αγοράς. Τέλος. Απλώς να το επαναλάβω γιατί άκουσα το επικρατικό σχόλιο της ε, Σιλβή ότι θέλω να παρουσιάσω αυτή τη μεταρρύθμιση υπό το του μανιχαϊσμού. Είναι πολύ εύκολο να το πούμε και αυτό και να λέμε ότι... Έχει να κάνει με το με το έργο από οι αποχρώσεις, χίλιες αποχρώσεις του Γκρι. Είναι πολύ εύκολο να το πει κανείς αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς ακριβώς οι, ε, δραστηριότητες των τραπεζών λιανικής μπορεί να ρυθμιστούν και αυτό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι να υποδοτούμε τις ε, χρημα... το οικονομικές ε, δραστηριότητες των τραπεζών με δημόσιο χρήμα. Σήμερα ε, συζήτησα με έναν από τους βασικούς ε, λομπίστες της ε, Deutsche Bank Και κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει εδώ στο Κοινοβούλιο και ένας υπεύθυνο του Βρετανικού ε, Υπουργείου ήταν εδώ και ζήτησε να μας πει ο κύριος Ρόκτο το εξής. Θα δεχόσασταν εφ' εξής η Deutsche Bank να χρηματοδοτεί τις ε, δραστηριότητε της στην αγορά με τις τιμές της αγοράς, δηλαδή χωρίς το πλεονέκτημα των κρατικών ε, ενισχύσεων. Ο κύριος απάντησε στην ερώτηση, όχι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για την Deutsche Bank ήταν απαράδεκτο να μην διαθέτει πλέον αυτήν την ε, κρατική ενίσχυση. Εν τω μεταξύ βεβαίως απολύθηκε ο άνθρωπος και καλά έκανε, αλλά ε, εάν ήταν ακόμη υπάλληλο, υπάλληλο της Deutsche Bank, τότε ήταν που θα τον πίστευα σε καμία περίπτωση. Αυτά λοιπόν να πω, νομίζω θα έχουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ακόμη και με το Συμβούλιο απέναντί μας, δεν ε, θα έλεγα ότι το Κοινοβούλιο με μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία θα πρέπει να θυσιάσει τις φοροδεξίες του και να τις φέρει στο επίπεδο των φιλοδοξιών του Συμβουλίου. Σκαζίλα μου ποιο το επίπεδο των φιλοδοξιών του Συμβουλίου. Κάτι άλλο που συνέβη χθε είναι ότι έδωσε το πράσινο φω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση των αποτελεσμάτων αναχώρα των διατάξεων του ΕΜΕΡ και του CRD4, λέγοντα ότι οι διατάξει αυτέ δεν θα είναι επιβλαβείς για την οικονομία. Επ' αυτού ε, το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε ομοφόνο και σχεδόν το ίδιο και το Συμβούλιο, διότι μόνο ένα κράτο μέλο συμφωνούσε με την άποψη του Κοινοβουλίου και 26 το αντίθετο. Τελικά υπερίσχυσε η δική μα η άποψη. Είναι λοιπόν και θέμα πολιτική βούληση. Εάν έχουμε πλειοψηφία και έχουμε ένα υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών, εάν κυρίε και κύριοι, κυρίω κύριοι Υπουργοί Οικονομικών, οι κύριοι μάλλον Υπουργοί Οικονομικών δεν βλέπουμε, δεν θέλουν να πάνε προ αυτήν την κατεύθυνση, δεν ξέρω γιατί θα του διευκολύνουμε το βίο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε Φιλίπ και τώρα Κατ Οκτώ ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Θα κλείσω τώρα τον κατάλογο και θα δώσω δύο λεπτά στον καθένα. Ο κύριος Μπάλτς πρώτος. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά ήδη αναφέρθηκαν λεπτομερώς. Εγώ δεν θέλω να μπω στην συζήτηση, ούτως ή άλλως δύο λεπτά έχω μόνο. Θα ήθελα να αναφέρω δύο γενικές σκέψεις θεωρώ πως ε, με την ε, Τραπεζική Ένωση που δημιουργήσαμε τον Απρίλιο πραγματικά πετύχαμε πολλά και τελικά συμφωνούμε όλοι με αυτό ε, θα συνεισφέρει στην οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη η Τραπεζική Ένωση και επίσης κάτι άλλο είναι σαφές. Η εφαρμογή της Τραπεζικής Ένωσης θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να σκεφτούμε τι συνολικά ε, ε έχουμε παραχωρήσει θα έλεγα στις, ε, στις εταιρείε που ε, δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών. Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να το συζητήσουμε και να δούμε ακριβώς το τι προτείνει η πρόταση της Κομισιόν. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποτε. Τέλος, η δεύτερη μου σκέψη. Το πρόβλημα και τα θέματα τα οποία αναφέρονται στην πρόταση της Κομισιόν οπωσδήποτε θα, αναφε... θα αντιμετωπιστούν από την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε πάντα το πρόβλημα too big to fail ή too big to save ή too complex to resolve. Επίσης ε, Σημαντικό είναι και αυτό το οποίο είπε ο Γκουναρ η προϋπόθεση για τις ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις των τραπεζών ε, οι προϋποθέσεις έχουν αλλάξει. Και το ίδιο πρέπει να γίνει και με την πρόταση της Κομισιόν. Εδώ πέρα λοιπόν σημαντικό είναι το μέτρο να διατηρηθεί. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για τις συζητήσεις ε, και αναμένω τις συζητήσεις που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Αυτό το οποίο θα επιθυμούσα εγώ είναι να κάνουμε κάπες να έχουμε κάποια ε, λιγότερα ρακτικόλεξα γιατί πραγματικά όλα αυτά τα αρχικά φτάνουν είναι κάπως υπερβολικά μάλιστα όχι η BRS λοιπόν ευχαριστώ Ελίζα Φερέιρα Παρακαλώ να μείνετε εδώ στον δύο λεπτών, γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα προσπαθήσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο τώρα συζητάμε. Αλλά το μικρόφωνο σας λέει ο γιατί δεν το έχει ανοίξει η ομιλήτρια. Νομίζω ότι πρόκειται για πολύ σημαντικό ζήτημα. Και θεωρώ ότι έχουμε όντως ε, κάνει πολλά μέχρι τώρα, αλλά τώρα πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι του ψηφιδωτού, κάτι το οποίο εκρεμεί πολύ καιρό. Και ο κίνδυνος είναι να μην μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε νομοθετήσει. Εάν ε, τις τεράστιες αυτές τράπεζες που είναι τόσο περίπλοκες, ε, αν τις, ε, τις αφήσουμε Χωρί κάποια δική προσέγγιση, μια που τόσο δύσκολο τις καταλάβουμε και να τις ελέγξουμε, να καταφέρουμε να τις κάνουμε ε, πιο ξεκάθαρε, ξεκάθαρες, πιο, πιο ε, επιδεικτικές ελέγχου με την νομοθεσία. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και αυτό το οποίο είπαν οι δύο-τρεις ε, συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο. Επίσης δεν ενεργούμε εν κενό. Υπάρχει μια σειρά πρωτοβουλειών στις ε, ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά σε Γερμανία επίσης και σε Γαλλία. Άρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα πρέπει το... σε ευρωπαϊκό πλαίσιο να οργανώσουμε τις τράπεζες και να οργανώσουμε μια τέτοια δομή, ούτω ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα συμφέροντα των πολιτών, των φορολογουμένων, να εξασφαλίσουμε μια ε, σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού σύστηματος στην Ευρώπη. Να μην γύρει πλάστιγκα υπέρ κανενός. ήδη κάποια κρατημέλη έχουν αρχίσει να βαδίζουν προς την κατεύθυνση. Επομένως, με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε την ε, προβληματική αυτή. Νομίζω ότι ήδη υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, το σωστό πνεύμα στο οποίο να κινηθούμε. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Τα Γιάννη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινώ από την παρατήρηση του Χόκμαρκ για τα 200 εκατομμύρια ευρώ που δεν έχουν επενδυθεί στην Ευρώπη και το θέμα και της πραγματικής οικονομίας που έθιξε ο κ. Λάμπερτς. Εάν μπλοκάρουμε την πραγματική οικονομία, εκεί θα εμποδίσουμε και τη χρηματοπιστωτική δράση. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να ξαναδώσουμε εμπιστοσύνη στους ε, δρόντες στην πραγματική οικονομία. Όχι με πολιτική παρέμβαση και υπερβολικούς κανόνες, αλλά με σωστού κανόνες δηλαδή. Θέλουμε ποιότητα. Αυτό που είπε και ο κ. Μπάλτ. Περισσότερη συγκέντρωση στην ποιότητα. Εμπιστοσύνη στου επενδυτέ. Διότι ο κίνδυνο είναι οι Ευρωπαίοι επενδυτέ να επενδύσουν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλε τι ε, ε, συναντήσεις που είχαμε τον κύριο Ρολέ, τον κύριο Ξαριέ Ρολέ, μου είπε ότι τα χρήματα υπάρχουν, τα χρηματοπροστατικά μέτρα υπάρχουν αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Οπότε δεν γίνονται και επενδύσει. Για να γίνουν σωστέ επενδύσει, χρειαζόμαστε και κανόνε που θα επιτρέπουν στι τράπεζε να λειτουργούν εντό τη πραγματική οικονομία. Και η πραγματική οικονομία δεν είναι μόνο οι τεράστιε επιχειρήσει, αλλά και οι μικρομεσαίε. Και εδώ ήταν σωστή επιλογή του Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια να προτείνει στη Βασιλεία 3 τον ε, παράγοντα στήριξη των μικρομεσαίων. Δηλαδή την πρόσβαση στι πιστώσει των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μιλάμε για πραγματική οικονομία και στήριξη τη πραγματική οικονομία, πρέπει να διακρίνουμε και μεταξύ μεγάλων ε, διεθνών τραπεζών και των μικρών οι οποίε πρέπει να προστατευτούν και από τα νέα κείμενα και του κανόνες που πρόκειται να εγκρίνουμε, διότι συχνά στηρίζουμε τελικώς ε, τους μεγάλους τραπεζικούς ομίλους και δεν κάνουμε αρκετά για να βοηθήσουμε τις μικρές. Τις μικρές που όμως ε, απευθείας ε, βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιτρέπουν την πρόσβαση στις πιστώσεις των οικογενειών. Οι μεγάλες τράπεζες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχει και ένα σύστημα κυρώσεων από τις ΗΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποια για τη λάθος διαχείριση του ε, ισοζυγίου τους. Και ήδη πρέπει να γίνουν κάποιες σχετικές προβλέψεις και τα απαραίτητα αποθεματικά. Αλλά να σκεφτούμε την πραγματική οικονομία πάνω απ' όλα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εκείνες θα στηρίξουν την πραγματική οικονομία ακριβώς. Και μετά περιμένουμε και την αγραμματότηση της Ήτρε ώστε να μπορέσει ο Χόκμαρκ να δουλέψει και να συμπεριλάβει στο κείμενό του μια απευθεία μνήα και επειδή είμαι συγκεκριτής από την Ήτρε θα κάνω ό,τι μπορώ και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση ε, να υπάρξει μια σχετική μνήα διότι συμφωνώ απολύτως με τον, Λάμπερτ, ε, με τον κύριο Λάμπερτ. Αν δεν υπάρξει ε, πρόσληψη προς την πραγματική οικονομία δεν μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα ούτε μακροοικονομικός. Ευχαριστούμε κυρία Νίνα Γκίλ από τους και δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να πω ότι με κάλυψαν πολλά από τα σχόλια που ήδη έγιναν. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, διότι στο παρελθόν όντως δεν το επιλύσαμε και νομίζω ότι γενικώ και η κοινή γνώμη δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη. Δεν πιστεύει ότι οι τράπεζες θα αυτορυθμιστούν. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα ζητήματα και να τα αντιμετωπίσουμε εδώ. Τα βασικά σημεία με τα οποία θα συμφωνήσω είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επιδοτούμε, να χρηματοδοτούμε τις τεράστιες αυτές που είναι too big to fail τράπεζες. Πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να πάνε παραπέρα. Κατά τη δική μου όμως άποψη δεν θα είχε νόημα αυτός ο κανονισμός αν δεν αντιμετωπίσουμε και τη σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα, την παράλληλη τραπεζική δραστηριότητα. Διότι Εάν το δει αυτό ε, και δείτε και τους αριθμούς που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο της Δημοσιονομικής Σταθερότητας, η παράλληλη τραπεζική δραστηριότητα είναι όσο ε, είχε τον ίδιο όγκο που είχε και πριν από την κρίση. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και για, επειδή είμαι η υπεύθυνη συγγήτρια για τα μέσα της, των χρηματαγορών, θα πρέπει και αυτό το θέμα να το λάβουμε υπόψη. Να προσθέσω λοιπόν τη φωνή μου σε αυτούς που είπαν ότι το βασικό σημείο της νομοθεσίας αυτής είναι να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την πραγματική οικονομία. Αυτό για μένα είναι το πλέον σημαντικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολντ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Εξεπλάγει από κάποιες από τις παρεμβάσεις ως τώρα αλλά νομίζω ότι η συζήτηση γενικώ πάει προς τη σωστή κατεύθυνση στην Ευρώπη. Επιλέξαμε μια σαφή αρχή για να διαθετήσουμε τα πράγματα. Με μια οικονομία κοινωνικού χαρακτήρα. Εδώ βλέπω οι παρεμβάσει να έρχονται από τα κόμματα που αυτές τις αρχές ακριβώς είχαν προωθήσει τελικά να μην τις ε, δέχονται και να μην είχαν τότε καθόλου κριτήρια για το πώς θα υποτιμήσουμε αυτό το νομοθέτημα. Η οικονομία της αγοράς όμως σημαίνει ανταγωνισμό. Κάποιες φορές έχουμε τέτοιους παράγοντες της αγορές που μπορεί να ασκήσουν την εξουσία τους σε μικρότερα κομμάτια της αγοράς. Αυτά τα μικρότερα λοιπόν κομμάτια της αγοράς πρέπει να δούμε πώς ορισμένοι από τους δρόντες μπορεί να περιορίζουν τελικά την ίδια τον ανταγωνισμό. Επίσης μια κοινωνική οικονομία της αγοράς σημαίνει ε, ότι υπάρχουν, ε, δεν υπάρχουν επιδοτήσει. Ε, και ότι ο επενδυτής θα πρέπει να καλύψει το ε, τίμημα εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Στις τράπεζες ευτυχώς υπάρχουν εγγύησεις για τους καταθέτες, αλλά υπάρχει κίνδυνος αυτή η εξορισμού δημόσια εγγύηση για τις καταθέσεις να χρησιμοποιηθεί για να επιδοτήσει τελικά άλλες τραπεζικές δραστηριότητες. Άρα πρέπει να υπάρξει διασφάλιση το ότι η αρχή ε, της, του σωστού ισοζυγίου ε, ε, και δεν υπάρχουν επιδοτήσεις. Επίσης η κοινωνική ε, οικονομία της αγοράς βασίζεται και στις επιλογές. Επιλογές χωρίς σύγκρουση συμφερόντων όμως πώς γίνεται. Ε, μια από τις βασικές αρχές πίσω από, την, από τον νόμο Γκλαστίγκελ είναι ότι αυτοί που κατασκευάζουν τα χρηματοστατικά προϊόντα δεν μπορούν να τα πουλήσουν σε όσους δεν έχουν αρκετέ πληροφορίες. Όλες αυτές οι συζητήσεις έγιναν βάσει της έκθεσης Λίκανεν και πραγματικά πλήσωμε που ελάχιστοι θυμηθήκαμε αυτή την έκθεση. Ο Λίκανεν τα ε, είχε θέσει αυτά ε, στις εξ αρχής. Ας μην παραβλέπουμε ότι έχει γίνει διεξοδική μελέτη των θέματων αυτών. Δυστυχώς δεν είχε συζητηθεί σύγκρουση συμφερόντων στην έκθεση εκείνη. Δεν τα είχε καλύψει αυτά. Αλλά αυτό που μπορούμε να μάθουμε από την έκθεση Λικάνεν είναι ότι αυτά δεν μπορούμε να τα κρίνουμε βάσει των γενικών αρχών, περισσότερων λιγότερων επενδύσεων, γενικών αρχών του εάν έχουμε κάνει πολλά ή λίγα, αλλά το ερώτημα είναι οι αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς τελικά έχουν γίνει σεβαστές τα τραπεζικά όπως σε άλλους τομείς. Πολύ φοβούμε ότι έχουμε έλλειψη σεβασμού των αρχών της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και μας σύρουν οι εθνικές προτεραιότητες για να σωθούν συγκεκριμένες κατηγορίες τραπεζών, κάτι που είναι τελείως αντιπαραγωγικό. Ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Χόκμαρκ που έχει καθορίσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να δούμε το όλο θέμα. Νομίζω φτάνουμε σε ένα χρονικό σημείο που με αυτό το πρώτο κείμενο που πρέπει να συζητήσουμε θα περάσουμε σε μια τεράστια συζήτηση, δηλαδή το πώς χρηματοδοτείται και προφοδοτείται η πραγματική οικονομία. Και από τις δύο όχθες του Ατλαντικού, ο τρόπος που οι δυναμικές αυτές σχέσεις ε, ε, συνδυάζονται για να δούμε εάν θα χρηματοδοτηθεί πρώτα η πραγματική οικονομία ή η παράλληλη, ε, κάτι που έγινε στι ΗΠΑ, ή εάν όπω εδώ θα ασχοληθούμε περισσότερο με τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ε, είναι και αυτό μια πρόπτικη και ταυτόχρονα ξεκίνησαν και διαπραγματεύσει για το TTIP, τη διατλαντική δηλαδή εταιρική σχέση, που μπορεί να επηρεάσει και την προσέγγιση μας αυτή την νομοθεσία ακόμα και αν θεωρούμε ότι το θέμα των προστατικών αγορών δεν θα συμπεριληφθεί. Στι ε, διαπραγματεύσει TTIP. Πέραν αυτού, νομίζω ότι το ευρωπαϊκό το οποίο έχει εξελιχθεί πολύ σε σχέση με το πότε ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση για το μέλλον τη διάθεση των τραπεζών. Μπορούμε να πούμε ότι με τη θέση σε ισχύ της Τραπεζικής Ένωσης σίγουρα θα επηρεαστεί η υγεία των τραπεζών ο αντίκτυπος αυτός δεν είναι ακόμη γνωστός σήμερα. Επίσης, τρίτο είδος σχολείου, νομίζω ότι σε σχέση με την πρόκληση της εσωτερικής αγοράς έχουμε ένα πραγματικό πρόβλημα μπροστά μας. Πρώτα απ' όλα το θέμα της διάρθρωσης των τραπεζών πρέπει να εξεταστεί ε, τμήμα ανά τμήμα ή με βάση τις κατηγορίες των τραπεζών και ανάλογα με την συμβολή του στη χρηματοδότηση, την τροφοδοσία τη πραγματική αγορά. Νομίζω ότι το να δούμε μία κατηγορία τραπεζών ή ένα είδο τραπεζική διοργάνωση καταλήγει σε μία τμηματική αντίληψη του πώς λειτουργεί η οικονομία αντιληψη του πω λειτουργει η οικονομια βασει των τραπεζών. Θα θυμάστε, κύριε Χόκμαρκ, τι κάναμε με την έκθεση Κάρας ε, στην περίπτωση της Επιτροπής Κρίσης. Αλλά να μην φτάσουμε σε κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς, σε κρατικοποίηση των διαφόρων ε, διαδικασιών, επανεθνικοποίηση δηλαδή, και να μην πετύχουμε το στόχο μας να αναβιώσει πλέον η ευρωπαϊκή οικονομία. Δύο συμπληρωματικέ παρατηρήσεις. Πρώτον, ότι τη συζήτηση αυτή, ο τρόπος που οι Ευρωπαίοι συμπεριφέρονται θα πρέπει να συζητηθεί και με βάση τη Βασιλεία και Στη συζήτηση αυτή κανείς δεν προτείνει ένα καλό deal, μια καλή συμφωνία στον τραπεζικό κλάδο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς αφού τμήμα ανά τμήμα, νομοθέτημα ανά νομοθέτημα θα έχουμε δει τις προκλήσεις της σταθερότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, τότε οι τράπεζες θα ξανασυμβάλλουν στη χρηματοδότηση της πραγματική οικονομίας. Ευχαριστώ. Σας ζητώ να παραμένετε στα χρονικά όρια παρόλα αυτά. Ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα προσεκτικά την όλη συζήτηση και έχω την αίσθηση πως στην έκθεση αυτή έχουμε de facto μια ανάλυση της ε, τρέχουσας νομοθεσίας ε, των ε, στόχων της νομοθεσίας της τραπεζικής δομής και θεωρώ πως η έκθεση αυτή είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία γιατί δεν κάνουμε μια γενική συζήτηση αλλά ξεκινάμε με αφετηρία την έκθεση Λικάνεν και την πρόταση της Κομισιόν και άρα αν λάβουμε υπόψη το τι έχει συμβεί από, ε, από το 2008 από τις ε, περιπτώσεις αυτές που ανέφερα και με τα too big to fail και τα ενσωματώσουμε εδώ θα έχουμε μια γενική έκθεση αξιολόγησης των ε, χρηματαγορών αλλά ακούσαμε ήδη πως ε, θα υπάρξει και μια αξιολόγηση αντικτύπου της αξιολόγησης και θα υπάρξει και μια έκθεση για το επενδυτικό πακέτο. Υπάρχουν λοιπόν τόσες πολλές εκθέσεις που δεν τις βλέπουμε όμως χωριστά. Γι' αυτό πραγματικά προτείνω οι εισηγητές όλων αυτών των εκθέσεων να καθίσουν μαζί και να εξηγήσουν τι κάνουμε που η μία είναι νομοθετική έκθεση, η άλλη είναι έκθεση αξιολόγησης, γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε ακριβώς πού θα δώσουμε βάρος, γιατί αν κάνουμε σε κάθε έκθεση γενική συζήτηση δεν θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει. έχοντας ε, ως αφετηρία την κοινωνική οικονομία της αγοράς, ε, τον ρόλο των τραπεζικών δομών και βεβαίως να τα συνδέσουμε αυτά με την έκθεση Λικάνεν και να δούμε τι θα γίνει με τις πτυχές των άλλων εκθέσεων γιατί δεν μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε αυτήν εδώ την έκθεση. αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια διαρδρωτική μεταρρυθμίση των τραπεζών. Γιατί θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση συνολικά των τραπεζικών δομών μετά την ε, έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό ακριβώς ε, ζητάμε ε, εμείς να καθίσουν όλοι οι ε, εισηγητές μαζί και να δουν ποια είναι η ουσία της κάθε μίας έκθεσης. Ευχαριστώ. Όλε Λουτβίξον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στην πρόταση αυτή. Για να ελέγχουμε και τις ε, μεγαλύτερες ε, τράπεζες σύμφωνα με την διαδικασία Λικάνεν η Κομισιόν πρότεινε να βρούμε μια λογική ισορροπία και να εφαρμόζουμε λογικά τους ε, κανόνες και αυτό δεν πρέπει να ισχύει μόνο για τις μεγαλύτερες τράπεζες θεωρώ Επίσης ε, θεωρώ πως είναι θεωτικό πως υπάρχει η δυνατότητα να δούμε την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, να τη δουν δηλαδή οι εποπτικές αρχές. Και βεβαίως μακροπρόθεσμα θα πρέπει να ε, υπάρξει μια εκλογήκευση των δραστηριοτήτων και του όλου συστήματος. Σας ευχαριστώ Μάρκο Βάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο και να παραμείνω εντό των δύο λεπτών. Είναι η πρώτη μου θητεία εδώ. Το 2009 όταν ξέσπασε η κρίση βρισκόμουν όντως σε μια εμπορική τράπεζα και ασχολούμουν με ποταμιεύσεις σε ένα κανονικό γκισέ και εγώ. Ελπίζω λοιπόν να μπορώ κάτι να συμβάλλω και εγώ γιατί όντως η κρίση που αντιμετωπίσαμε ήταν συστημική. Άκουσα τον εισηγητή που είπε ότι πολλά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια Όντω πολλά έχουν γίνει, αλλά με ποιο σκοπό, τι άλλαξε. Αυτό που ίσω άλλαξε είναι ότι οι επιχειρήσει, αυτέ που ασχολούνται περισσότερο με την πραγματική οικονομία και ο παραδοσιακό τραπεζικό κλάδο, αυτέ που ουσιαστικά προάγουν το ΑΕΠ, την απασχόληση και τι θέσει εργασία, αυτέ ε, πτώχευσαν. Και όλη η, πραγματική, η συστημική πραγματικότητα, οι μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε, αυτέ που ασχολούνται με μεγάλε ε, δράσεις και συναλλαγές, αυτές είναι που στηρίχθηκαν από τις κεντρικές τράπεζες, τις εθνικές τράπεζες, με, ένα, με μια κατεύθυνση που πήρε το όλο τραπεζικό κύκλωμα πολύ λανθασμένη. Εδώ λοιπόν κάτι θα πρέπει να κάνουμε, λέμε, για να δώσουμε τέρμα σε αυτή την κρίση. Μα πώς τις τραπεζικές υπηρεσίες θα τις κάνουμε να λειτουργούν προς όφελος της πραγματικής οικονομίας και να προάγουμε αυτά που λέμε τώρα, την απασχόληση, την ε, επαναδιανομή του πλούτου Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακριβώς πρέπει να αναζητήσουμε με εντατικές προσπάθειες στην, μετά την αποστήρωση ε, και όχι να κάνουμε μια μικρή ανώδυνη παρέμβαση, αλλά κάτι πολύ ε, έντονο και ριζοσπαστικό. Να κάτσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να εργαστούμε σοβαρά και να προσπαθήσουμε να αποστηρώσουμε, να, να να σπάσουμε μάλλον το απόστημα της κατάστασης αυτής. Ε, της κατάστασης στην πραγματική οικονομία που επηρεάζεται και από τη διεθνή πραγματικότητα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο τώρα στον εισηγητή, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή, τους σκιώδους εισηγητές και όλους όσοι έλαβαν τον λόγο. Ήταν πολύ χρήσιμο όσα ακούσαμε σύντομα να σας ε, επισημάνουμε τρία τεινά. Πρώτα-πρώτα γιατί χρειαζόμαστε μια μεταρρύθμιση μετά από όλες τις άλλες που προηγήθηκαν. Δεν θέλω να φοβήσω τον κύριο Μπάλτς με ε, όλα αυτά τα αρχικά, αλλά τέλος πάντων έχουμε ε, ε, το καινούριο πλαίσιο για την κεφαλοχή επάρκεια, αλλά αυτό δεν είναι πανάκια. Είπε η ανάλυση ότι όταν δούμε την πολιτική των τραπεζών βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε σχέση με το πώς παίζουν τους κινδύνους ε, και είδαμε ότι δεν επαρκεί τα τη κεφαλής επάρκειας τόσο έχουμε κάνει μέχρι τώρα, επομένως είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι το φάρμακο για όλα. Οπότε όσον αφορά το τι κάναμε για τις τράπεζες, θεωρούμε ότι αυτό το νομοθέτημα είναι επαργέστατο. Όμως, μερικές από αυτές τις περίπλοκες, τις πολύ μεγάλες τράπεζες που σχεδιάζουμε για αυτό το, που συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, ε, αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση. Και επομένως, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για αυτές τις τράπεζες που, ζουν, που δρούν διασυνοριακά. Υπάρχει επομένως πάντοτε κάποιο κίνδυνο τον οποίο διατρέχουν και αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Επίση, ε, έχουμε τη διάσταση ιστορική αγορά και συμφωνούμε ότι αυτή η διάσταση ήταν πολύ σημαντική. Ε, ήδη κάποια κράτη-μέλη έχουν νομοθετήσει σχετικά και άλλα ε, μελετούν ε, το να γίνει τέτοιου είδους νομοθεσία όσο δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νομοθετήμα. Αλλά εκτός από την ενιαία αγορά ε, έχουμε και το ότι αυτού του είδους η απόκληση των εθνικών νομοθεσιών είναι ένας κίνδυνος και ένας πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης είναι αυτό το ενιαίο εγχειρίδιο που το οποίο δεν πρέπει με άστοχη νομοθεσία να το υπονομεύσουμε. Δεν είμαστε κατά των ε, παγκοσμίων τραπεζών. Δεν θέλουμε να μην συγκροτηθούν τέτοιοι όμιλοι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος των κινδύνων, να περιοριστούν στο αποδεκτό επίπεδο. Δεν θέλουμε η πραγματική οικονομία να δυναμητίζεται, να υπάρξει συμπληρωματική προσπάθεια μεταξύ εθνικής νομοθεσίας και κοινοτικής και όλοι οι εμπλεκόμενοι να μπορούν να σταθούν στην Τραπεζική Ένωση. Τα είπε η κυρία Γκουλάρ, τι γίνεται με το Συμβούλιο, ιδίω όσον αφορά την διακριτική ευχαίρεια για την εποπτεία. Α, όμως ε, δεν είναι ομόφωνο το Συμβούλιο σε αυτό. Ακόμα γίνονται ζημώσεις εκεί για να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν. Εμείς έχουμε την πρότασή μας που θεωρώ ότι είναι ρεαλιστική και προσπαθούμε οι υποπτικές αρχές να έχουν μέχρι ενός σημείου ευελιξία και διακριτική ευχέρεια στις ενέργειές τους, κάτι το οποίο είναι ρεαλιστικό, γιατί είναι περίπλοκος ο κόσμο που ζούμε. Ε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Και τώρα, τελευταίο λόγο, ο εισηγητή μα, ο Χόκμαρτ. ευχαριστώ πολύ. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και μου άρεσε πάρα πολύ το ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι από την αριστερά ε, τοποθετήθηκαν σαν ε, πραγματικοί καπιταλιστέ τη οικονομία τη αγορά. Ε, αγοράς. Πολύ καλή αφετηρία αυτή, πολύ καλή βάση συνεργασία. Δηλαδή συμφωνείτε μαζί μα. Δεν και Ισλάμ. Ε, ναι, πάντοτε, πάντοτε όταν το πάνε καλά τα πράγματα. Βεβαίω, η κοινωνική οικονομία της αγοράς, συμφωνούμε. Και εσείς ελπίζω συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις. Ο Ότμαρ είπε κάτι πάρα πολύ σωστό, το οποίο θα πρέπει να μην το ξεχνούμε για τα συμπράσματα που θα εξαγάγουμε ότι μιλάμε τώρα μόνο για ένα από τα πρόνομο θετήματα που χρειάζονται. Μόνο ένα κομμάτι του ψηφιδωτού. Πολλές φορές είναι σωστό να τα λέμε όλα. Γιατί κάποιος νομίζω ο Φιλίπ το είπε. Είπε κάτι για μουσική και συμφωνώ μαζί του. Αλλά πολλές φορές αλλάζει ο σκοπός. Δηλαδή, να δούμε τι γίνεται με, το, με την πολυνομία. Από το 2009 έχουμε βγάλει ένα νομοθετήματα. Δεν είπα εγώ ότι αυτά είναι προβολικά πολλά. Είμαι ευχαριστημένος και νομίζω ότι έτσι αλλάξαμε το τοπίο. Εμένα αφετηρία μου είναι το ότι το 2014 είναι τελείως διαφορετικό από το 2009. Άλλαξαν όλα. Και αν κανείς έχει σεβασμό και νομίζω ότι εμείς έχουμε, θα πρέπει να αποδεχθεί το ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με όταν ξεκινήσαμε αυτή την διαδρομή. Η νομοθεσία αυτή δεν θα πρέπει να θεωρείται κάτι το αυτόνομο, ανεξάρτητο από όλα τα άλλα, ούτε είπα. Όπως είπε ο Σάιτ Καμάλ, ο φίλος Καμάλ, ότι προτιμώ ότι σε αυτές τις ε, παγκόσμιες τράπεζες. Ή όπως είπε ε, κάποιος ε, φίλος από την κέντρο αριστερά ότι μου αρέσουν οι τράπεζες. Όχι, όχι, όχι, προτιμώ να αγαπάω πρόσωπα και όχι φορείς. Αλλά θέλω να υπάρχει εκεί πολυμορφία, να αντιστοιχεί στην ε, ζήτηση. Έχουμε λιανική, λιανικές υπηρεσίες, έχουμε επενδυτικές υπηρεσίες από τις τράπεζες κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει τέτοιου είδου ροή και εξέλιξη. Δεν θέλω οι λιανικές υπηρεσίες να απομονώνονται από την πολιτική ρευστότητα και το λέω αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Περί αυτού πρόκειται. Να δούμε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Είδαμε ποια είναι τα προβλήματα όσον αφορά τι επενδυτικέ τράπεζε. Και βρίσκαμε το πρόβλημα τη αντιπαράθεση ε, των ελληνικών υπηρεσιών με ε, τι θεραστικέ τράπεζε. Είδαμε τι έγινε με τη Lehman Brothers. Πολλέ φορέ αποτελεί παράδειγμα το τι γίνεται εκεί στη ΣΥΠΑ. Ότι αυτοί εισήγαγαν τα προβλήματα των λιανικών τραπεζικών υπηρεσιών σε σχέση με, τη, με την αγορά τη στεγαστική. Οπότε αυτή την αντιπαράθεση των δύο κατηγοριών υπηρεσιών ή τραπεζών. Άρα αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε οπότε και τότε θα μπορέσουμε να δούμε και τα προβλήματα τα σχετικά με το trading και την κερδοσκοπία. Θα πρέπει πολλές φορές να είμαστε ομοί αλλά ομοί και σκληροί σε σχέση με τα πραγματικά προβλήματα. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των κινδύνων, όπως είπε η Κομισιόν, ότι δηλαδή οι παγκοσμίες τράπεζες μπορούν να μας οδηγήσουν σε τέτοια κατάσταση, αλλά να το δούμε αυτό έχοντας υπόψη όλο το υπόλοιπο ψηφίδωτο, όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα τα οποία ήδη έχουμε θεσπίσει. Είναι διαφοροποιημένες οι κεφαλογικές απαιτήσει. Αυτή η οδηγία για την κεφαλογική επάρκεια σε αυτό αφορά. Στη διαφοροποιημένη αντιμετώπιση. Το BDRD. Πολλές φορές λέμε ότι μπορεί μεγάλες για να πτωχεύσουν κάποιες τράπεζες κλπ. Σημαντικό αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρξουν. Θα πρέπει επομένως να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι κανόνες, η νομοθεσία, ό,τι χρειάζονται αυτές οι τράπεζες. Τέλος, για τις επιδοτήσεις. Ευχαρίστως όλα αυτά να τα συζητήσουμε και διμερώς, εκτός από την Επιτροπή. Εάν θέλουμε, να εξασφαλίσουμε την αντίδρασή μας με το που ξεκινάνε προβλήματα ε, για κάποια τράπεζα και να μην προσφεύγουμε αμέσως στα χρήματα των φορολογουμένων, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη αυτή τη δομή που προβλέπεται όσον αφορά ε, την σωτηρία των τραπεζών ότι όλα αυτά που έχουμε θεσπίσει να αποδίδουν. και να υπάρχει και διαφοροποίηση στη γεωβολική επάρκεια της τράπεζας, στα τέλο πάντων στο ενεργητικό της. Ας πούμε, τράπεζα ελληνικών τραπεζικών εργασιών, αν ήταν μόνο τέτοιες οι τράπεζες με τις οποίες ασχολούμαι θα έχω το πολύ καιρό. Ε, τότε δεν θα είχε αξιοπιστία η ισοτερία της τράπεζας με ίδια μέσα, τον Μπέιλιν. Ε, γιατί τότε θα βρεθούμε στην, στη συνταγή σωτηρίας μέσω των καταθετών όπως έγινε στην Κύπρο. Να η κοινωνική διάσταση που είπατε. Όλα αυτά υποσκάπτουν, υπονομεύουν την αξιοπιστία. Άρα, να μην δούμε τα πράγματα ιδεαλιστικά. Αλλά πιο ασφαλή είναι τελικά οι τράπεζες λιανικής. Όμως, έχουμε μεγάλη ποικιλία τραπεζών και άρα έχουμε ποικιλία κινδύνων και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να, ποια είναι η αφετηρία. Πρέπει να υιοθετήσουμε γιατί σίγουρα αγαπητοί φίλοι φίλοι και Σβέν που είστε εραστές της οικονομίας της αγοράς. Αν είχαμε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση και είχαμε τα χρήματα των καθετών σε σε κάποιες ε, από αυτές τις ε, τοπικές ε, τράπεζες λιανικής και κινδυνευαν οι καταθέσεις. Τι θα λέγατε, είμαι σίγουρος ότι θα λέγατε όχι, όχι, σωτηρία, σωτηρία με ίδια μέσα. Δεν ξέρω. Θα είχατε το κουράγιο. Έχετε κουράγιο για άλλα πράγματα, Φιλίπ, και σας θαυμάζω. Γκούναρ, σε ευχαριστώ, λέει ο Φιλίπ. Λαμπέρ, η πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκεται δεν έχει το κουράγιο να κάνει αυτέ τι κινήσεις. Αυτό σημαίνει δεν το έχουν και οι άλλοι. Νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να αναλαμβάνει και τις, ε, τις συνέπειες. Νομίζω ότι κάθε απόφαση μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή, γιατί και αυτό και εγκατακλείδει αυτό τελικά, κύριε Πρόεδρε, αυτό και προτιμώ. Δηλαδή, όταν μια τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα, προτιμώ ο καπιταλιστής που εσείς λατρεύετε να πληρώσει την ύφη και να είναι ασφαλής η καταθέτες. Να τι πάει να πει κοινωνική, σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το στόχο, αλλά διαφέρουμε όσον αφορά το μόνο πάτη που να ακολουθήσουμε. κοινωνική οικονομία της αγοράς. Αλλά τώρα μιλούμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χόγμαρκ, διακόπτη. Από σε ΕΛΚ, κύριε Πρόεδρε, είμαστε ευτυχείς τώρα που όλοι θέλουν οικονομία της αγοράς. Πρόεδρος. Ναι, ναι, υπάρχει ολόκληρη προβληματική για το κατά πόσο η ελεύθερη οικονομία της αγορά έχει κοινωνικό χαρακτήρα ή θα πρέπει να αποκτήσει κοινωνικό χαρακτήρα. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε πολλές διαφορετικές ε, απόψεις για το πώς θα αποκτήσει κοινωνικό χαρακτήρα η οικονομία της αγοράς, τέλος πάντων. Πρόκειται να κάνουμε την ε, σχετική ακρόαση στις 2 Και το σχέδιο της γνωμοδότησης θα προσφερθεί 21 Δευτέρου και η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 13 Πρώτου και θα μελετήσουμε τις τροπολογίες στις 23 Δευτέρου. Θα ψηφίσουμε 23 Τρίτο και στην Ολομέλεια του Απριλίου πρόκειται να κριθεί και ψηφιστεί η έκθεση. Αυτά για το τόσο ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Και τώρα προχωρούμε σε ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο έχει σχέση με αυτό που μόλις συζητήσαμε. Πρόκειται για μια δέσμη προτάσεων της Ευρωπαϊκής σε σχέση με την πρότασή μας του Ιανουαρίου του 2014 και πρόκειται για το σχέδιο εικονισμού όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότηση τίτλων. Ο κύριος Ρενάτο Σόρο είναι ο εισήγητης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως μόλις είπατε, Ο κανονισμός αυτός έρχεται ως μια δέσμη νομοθετημάτων στο Κοινοβούλιο μαζί με άλλα νομοθετήματα όπως αυτό που μόλις συζητήσαμε και με, το, με τρόπο τόσο ενδιαφέροντα και τόσο παθιασμένο για την μεταρρύθμιση, τη διαφορετική μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος. Και η διαφάνεια των συλλαγών χρηματοδότηση τίτλων προκύπτει και εμπνέεται από την έκθεση Λικάινεν το 2011. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, φτάνουν στα χέρια μας μαζί, διότι η... το σύστημα αυτό με την διασφάλιση των ε, τίτλων και της χρηματοδότησής τους καθώς και των σχετικών συναλλαγών με εγγυήσει, με τη σχετική κάλυψη των δανείων και του λεγόμενου θιόντος τραπεζικού τομέα πρέπει να καλυφθούν με κάποιες διατάξεις. Έχει προκύψει ο κίνδυνος ότι κάποιες ε, από τις κλασικές συναλλαγές του τραπεζικού συστήματος μπορεί να ξεφύγουν από αυτό το κλασικό τραπεζικό σύστημα για να πάνε στην ε, σκιώδη τραπεζική ε, δραστηριότητα. Το πρώτο που έκανα λοιπόν είναι ότι όταν ανέλαβα την έκθεση αυτή συζήτησα με τον συνάδελφο που μόλις έφυγε, τον Χόκμαρκ. Τον κύριο Χόκμαρκ. Όμως αυτό που θέλουμε με την όλη συζήτηση είναι να έχουν μια διαφορετική πορεία, παρόλο που θα συμβαδίσουν, τα δύο αυτά νομαθετήματα. Είχαμε ήδη άτυπη συνάντηση και συνομιλίες για να καταλάβουμε ποια μπορεί να είναι η συνεννόηση μεταξύ μας και αποφασίσαμε να ε, να έχουμε μια παράλληλη πορεία όπως προβλέπεται και για την πρόταση του κυρίου Χόκμαρκ. Σήμερα λοιπόν γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μέχρι τα Χριστούγεννα στις 18 Δεκεμβρίου θα υποβληθεί το πρωτοσχέδιο έκθεσης που θα συζητηθεί στην Επιτροπή στις 21 Ιανουαρίου. Στις 27 Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες και Εντός Μαρτίου ελπίζουμε το θέμα να φτάσει να ψηφιστεί στην Επιτροπή. Η διαφάνεια των συνελεγών χρηματοδότησης τίτλων αφορά την πώληση τίτλων ε, για σκοπούς ε, αγοράς και για να, ε, να μπορεί να δημιουργηθεί ρευστότητα για τον αγοράστη και τα δάνεια, το, τη διανεοδότηση τίτλων χωρίς την υποχρέωση επαναγοράς. Εδώ υπάρχει και η δυνατότητα rollover μετακύλησης που ε, παρατείνει την ε, διορία. Μιλάμε για ένα τεράστιο τομέα, 53, ε, 153 μάλλον 3 ευρώ που κάνουν την ευρωπαϊκή αγορά πρώτη στον κόσμο εδώ. Ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείες. Ένα μεγάλο κομμάτι βεβαίως βρίσκεται στην ε, Αγγλία, όπως ξέρουμε, που είναι μια μεγάλη χρηματοοικονομική και χρηματοπιστωτική αρένα. Με σκοπό σκοπό να μειωθεί, το συστημικό, να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος, το Financial Stability Board, το Συμβούλιο Δημοσιονομικού Κινδύνου, προέβλεψε κάποια κριτήρια για την προστασία της πώληση τίτλων με σκοπό την επαναγορά στα πλαίσια του σκιώδους τραπεζικού συστήματος. Εδώ ε, ε, αυτά που προτείνουμε εμείς ακολουθούν τις συστάσεις του ε, FSB ιδίως την υπαριθμόν δύο σύσταση, δηλαδή την υποχρέωση συλλογής στοιχείων για την χρηματοδότηση της αγοράς μέσω τίτλων και προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Η σύσταση επίσης υπαριθμόν 5 επιβάλλει στους εμπειρογευμένους να είναι ε, και ως προς τους επενδυτές τους διαφανείς και επίσης η σύσταση 7 που προβλέπει για τους ε, συνελασσόμενους να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στους πελάτες τους. Τρία επίπεδα λοιπόν ε, ενημέρωσης και πληροφόρησης στο συστημικό επίπεδο ως προς τους επενδυτές και μετά ως προς τους επιμέρους, τους μεμονωμένους πελάτες, ιδιώτες. Ο κανονισμό θέλει να δημιουργήσει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα πιο σταθερό και πιο ασφαλέ, με διατάξει που έχουν να, να ε, βελτιώσουν, να αυξήσουν τη διαφάνεια στα τρία αυτά επίπεδα. Η συμβατική διαφάνεια είναι εξίσου σημαντική, όχι μόνο εναντί των επενδυτών, διότι οι διάφοροι τίτλοι όχι απλώ χρησιμοποιούνται για την δημιουργία ρευστότητα, αλλά πολλέ φορέ στη συνέχεια ε, ξαναχρησιμοποιούνται για περαιτέρω δημιουργία ρευστότητα. Δημιουργείται λοιπόν έτσι ένα πύργο, μια πυραμίδα ε, Κάποιε φορέ κάποιοι από αυτού του τίτλου χρησιμοποιούνται και 10 φορέ. Άλλοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν 4 φορέ στη σχετική αγορά. Στην Ευρώπη δεν έχουμε ακόμη αυτέ τι πληροφορίε. Οι αριθμητικέ πληροφορίε ισχύουν για την Αμερικανική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εντωμεταξύ, λόγω τη σημασία του τομέα αυτού, ε, δήλωσε ότι ένα από του λόγου τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2009 είχε να κάνει με το υπερμεγέθες χρηματοπιστωτικό σύστημα που ήταν και πολύ χρεωμένο, ε, με μεγάλη έκθεση. Το να καταλάβουμε λοιπόν αυτήν την ε, επαναχρησιμοποίηση, να καταλάβουμε μάλλον πόσο είναι αυτή η έκθεση σημαντική και το κατά πόσο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό με την ε, διασφάλιση των χρηματοδότηση τίτλων είναι πολύ σημαντικό. Στι πρώτε μας συζητήσει με τους σκιώδη, με κάποιου προσώπου ευρωπαϊκών οργανισμών, με ενώσει και υπεύθυνου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και εκπροσώπου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και του Συμβουλίου Δημοσιονομικού Κινδύνου, προέκυψε η κοινή με έρημνα να προχωρήσει αυτό το νομοθέτημα. Φυσικά κάποια επικριτικά σχόλια παραμένουν. Κάποια λιγότερο ζωτική σημασία, κάποια ε, σημαντικά. Πρώτα απ' όλα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση τη ε, ορολογίας. Πρώτα απ' όλα μεταξύ των κρατών ε, μελών, αλλά και για να ευθυγραμμιστούμε και με τις υπόλοιπε αγορές, την Αμερικανική και τι Ασιατικέ ευθυγράμμιση λοιπόν ε, της ε, ορολογίας και των ορισμών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράστηκε υπέρ ε, υπέρ της χρήσης του όρου επαναχρησιμοποίηση, reuse και όχι rehypothecation, η επαναπόληση. Υπάρχουν δηλαδή πολλές δυνατότητες σε έναν τίτλο με τελικό σκοπό την πώληση για την επαναγορά. Υπάρχει και η περίπτωση της ε, δανειοδότησης. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή κανείς ένα προσωρινό ε, αποθεματικό που έχει στο χαρτοφυλάκιό του. Ακόμη πιο εύστοχο θα ήταν να ορίσουμε το πεδίο του νομοθετήματο σωστά. Δηλαδή, αν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε που σήμερα γνωρίζουμε και που ε, απαντώνται συχνά στην αγορά ή και για μελλοντικέ χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Νέε που μπορεί να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Τι χρηματοπιστωτικέ λοιπόν υπηρεσίες μπορεί να τις ε, συλλάβουν κάποιοι με τρόπο ώστε να παρακάμπτουν την νομοθεσία. Γι' αυτό πολλοί από τους ενδιαφερομένους, τους ε, εμπλεκομένου εδώ, θεωρούν ότι θα πρέπει η νομοθεσία αυτή να είναι αρκετά τα ευρεία αναθέτοντα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρόπο πολύ συγκεκριμένο να αναλάβει τη σωστή υλοποίηση για παρόμοιε συναλλαγέ στο μέλλον ακόμη και αν σήμερα δεν γνωρίζουμε το χαρακτήρα και το όνομά τους αλλά που θα μπορεί να του προβλέψουν οι συναλλασσόμενοι στο απότερο μέλλον. Ένα άλλο επικριτικό σχόλιο είναι το εάν στο νομοθέτημα αυτό θα πρέπει να εντάσσονται και κεντρικές τράπεζες. Διότι οι δράσεις ρήπο που τις ε, αναλαμβάνουν συνήθω οι κεντρικές τράπεζες έναντι των συναλλασσομένων ή των αντισυμβαλωμένων, ίσως και αυτές θα πρέπει προσωρινώς ή διμερώς να γνωστοποιούνται στις αρχές εποπτείας. Κάποιοι λένε ότι η νομοθεσία θα πρέπει να καλύπτει και τις κεντρικές τράπεζες και να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα ή όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Ε, μεταξύ το, αλλά άλλοι, ε, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θεωρεί ότι δεν μπορεί οι ίδιοι κανόνες να ισχύουν για τις κεντρικές τράπεζες που ε, θα σχεδιάζουν και την νομισματική πολιτική που πρέπει να είναι άμεση, πρέπει να είναι ε, έγκαιρη για να είναι αποτελεσματική. Θα είναι λοιπόν δύσκολο να είναι τόσο διαφανεί οι τράπεζε αυτέ ω προ την αγορά. Όμω το θέμα τη συμπερίληψη των κεντρικών τραπεζών είναι κάτι που ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί. Το συζητούμε. Κάποιε πολιτικέ ομάδε θεωρούν ότι ο κανόνα τη διαφάνεια θα πρέπει να αφορά να αφορά μόνο την νομισματική πολιτική που χαράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. ένα ακόμη θέμα που θα μπορούσε κανείς να μελετήσει περαιτέρω και μετά τη συνάντηση που είχαμε την υπεύθυνη της, ε, ε, από το Αμερικανικού Υπουργείου ήταν το αν θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το reporting αυτού του κλάδου με το reporting που γίνεται στην Αμερικανική αγορά συγκεκριμένα. Δηλαδή αυτή η διμερής καταγραφή να ε, συνδυαστεί με μία ε, κοινή αναφορά στις συναλλαγές και προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναλήψεις και επικαλύψεις. να αποφευθούν εκεί που τα στοιχεία ούτως ή άλλως αποκαλύπτονται, δημοσιοποιούνται. Όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν οι συγκεκριμένες τεχνικές που προβλέπει το ΕΜΙΡ. Δηλαδή το σύστημα καταγραφής των συναλλαγών για τα παράγωγα. Εδώ θα πρέπει να ορίσουμε τα σωστά πρότυπα για, την, ε, για το επίπεδο προστασία που θα προβλέψουμε στο σύστημα διαφάνειας συναλλαγών και χρηματοδότησης τίτλων. Θα πρέπει να βασιστούμε λοιπόν στα όσα προβλέπει το ΕΜΙΡ και τα πρόσφατα διδάγματα για να μην έχουμε τα ίδια σφάλματα με το παρελθόν. Επίσης υπάρχει το θέμα των κουρεμάτων των haircuts και αν θα πρέπει να ε, διευθετηθεί ή να προβλεφθεί ένα ελάχιστο όριο όπως έχει ζητηθεί για αυτές τις συναλλαγές είτε για να είναι μικρότερη κίνδυνη που αναλαμβάνει ένας μεμονωμένος ε, συναλλασσόμενος ή παράγοντας στην αγορά και που δανείζει χρήμα έναντι της προσωρινής ε, απόκτησης ή αγοράς τίτλων. Με συγχωρείς, ε, με συγχωρείς. αν μπορείς Ρενάτο να κλείσεις σε κανένα λεπτό, διότι μετά έχουμε να ακούσουμε και τους σκιώδεις. Εντάξει, ολοκλήρωσα. Το θέμα των haircuts λοιπόν συμπεριλαμβάνει έχει κινδύνους για τις μεμονωμένε τράπεζες αλλά και συστημικούς κινδύνους διότι θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί στο δινεκές ο αριθμός ε, και το πόσες φορές ένα συγκεκριμένο στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ρευστότητα μεν, αλλά με την πρόκληση τεράστιων κινδύνων κυρίως συστημικών. Εδώ έχει φτάσει όλη η συζήτησή μα. Ε, με μεγάλη χαρά θα ακούσω τα σχόλια των υπολείπων σκιωδών εισηγητών. Και αν υπομονώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση ή μεταξύ των σκιωδών. Ευχαριστώ. Renato, now the first... Ευχαριστώ Ρενάτο. Τώρα ο σκιωδής ή η σκιωδής του ΕΛΚ δεν τα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μια αναφορά σε αυτό το οποίο είπε ο Γκούναρ και τη σύγκριση του σήμερα με το 2009. Πράγματι είμαστε το 2014, αλλά έπρεπε οι κανόνες αυτοί να έχουν τεθεί πολύ νωρίτερα δεδομένης πλέον της ε, εμπειρίας μας. Αφενός πρόκειται για συναλλαγές που έχουν μεγάλη σημασία για την ρευστότητα της αγοράς, αλλά ταυτόχρονα είναι συναλλαγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο επικίνδυνο στον σκιώδη τραπεζικό τομέα για να ε, δημιουργηθεί υπερβολική μόχλευση με τον κίνδυνο μετάδοσης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο κανονισμός και ακριβώς αντιμετωπίζουμε εδώ πέρα δύο προκλήσεις. Η μία είναι το να συνεργαστούμε με τον Γκούναρ και τους κοιόδης ηγητές στην έκθεση Λικάνου και είναι σαφής η σύνδεση εδώ, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε πως ε, ίσως ε, θα μπορούσαμε να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα εδώ πέρα σε σχέση με την έκθεση Λικάνου. Πρέπει λοιπόν να δούμε σε ποιο βαθμό θα είμαστε συντονισμένοι ίσως κάποια στιγμή μπορεί να ληφθεί μια απόφαση για να μοιράσουμε τις δουλειές αλλά ταυτόχρονα εκ παραλλήλου στο πλαίσιο της σκιώδους τραπεζικής βλέπουμε πως γίνεται πάρα πολλή δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικά το Συμβούλιο δημοσιονομικής ε, σταθερότητας ε, κοιτάει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει επίσης η ιδέα της, ε, των ρήτρων, ανα, ρήτρων αναθεώρησης κτλ. Οπότε βρήκαμε κάποιους τομείς τους οποίους θεωρούμε πως θα ε, ήταν χρήσιμες κάποιες ε, τροπολογίες. Ε, ένας τομέας είναι βεβαίως οι ορισμοί. Ήδη το 2014 είμαστε σε θέση να πούμε πως πολλοί ορισμοί βρίσκονται σε άλλα νομοθετήματα και μπορούμε να έχουμε άρα μια ενιαία φιλοσοφία. Πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα υπάρχουν όπως sell by or buy, sell back transactions και τα λοιπά αλλά υπάρχουν βεβαίως και ορισμοί που μπορεί να απαιτούν κάποια μεγαλύτερη ακρίβεια στο πλαίσιο του κανονισμού αυτών. Οπότε είναι δύσκολο το ζήτημα αυτό και βεβαίως πάμε πολύ πέρα από τους ορισμούς, αλλά είναι και αυτό μία πρόκληση. Μετά. Το μεγάλο ζήτημα που επίσης αναφέρθηκε από τον Ρενάτο είναι το τι γίνεται στις καταστάσεις όπου μπλέκονται οι κεντρικές τράπεζες αντισυμβαλόμενοι και το εάν οι συναλλαγές αυτές θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στον κανονισμό ή όχι, τα ρέπος και τα λοιπά, οτιδήποτε συνδέεται με την νομισματική πολιτική. Μεγάλο ζήτημα και πράγματι μπορεί να υπάρξει κάποια εξαίρεση εδώ για τις συναλλαγές αντισυμβαλωμένων και των κεντρικών τραπεζών. Και ένα άλλο ζήτημα αφορά κάπως ε, τις απαιτήσει ε, ενημέρωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη. Και νομίζω πως είναι θεμητό να εξετάσουμε κάποιες εξαιρέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βεβαίως ε, τις συναλλαγές να τις δηλώνουν οι χρηματοπιστωτικοί αντισυμβαλόμενοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έτσι θα είναι μικρότερο το βάρος. Τώρα υπάρχει το ζήτημα του χρονικού περιθωρίου για το οποίο πρέπει να διατηρούν τα αρχεία των συναλλαγών ε, οι επιχειρήσεις. Ε, η πρόταση Κομισιόν είναι αρκετά γενναιόδορη φτάνει τα 10 χρόνια και βεβαίω μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ε, την περίοδο αυτή. Αν λάβουμε υπόψη τον δυναμισμό των αγορών και η δεκαετής περίοδος δεν έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε μία μικρότερη περίοδο. Υπάρχει επίσης γενικότερα το ζήτημα το εξή. αν θέλουμε να συνεισφέρει αποτελεσματικά ο χρηματοπιστωτικό τομέα στην ανάπτυξη, πρέπει να δούμε και το κόστος των νέων κανονισμών. Η διαφάνεια είναι απολύτως ουσιαστική σημασία, αλλά δεν έχω πιστεί πως χρειάζεται ο ίδιο βαθμό λεπτομέρειας από την πλευρά των ε, πολιτών και ε, ίσως ε, θα μπορούσε να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Και με αυτό το σκεπτικό, δηλαδή να μειώνουμε το κόστος των νέων απαιτήσεων για τις επενδύσεις, νομίζω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα εγκριστάμενα μέσα. Παραδείγματος χάρη, ε, τα διάφορα αποθετήρια θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για να μειωθεί το κόστος για τους επενδυτές και τέλος θεωρώ και το είπες Ρενάτο ανέφερες τα ρέπος και τη δουλειά που γίνεται στο Συμβούλιο Συστημικής Σταθερότητας, στο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας. Πραγματικά, απαιτούνται πολλές εγγυήσεις όταν ένα μη τραπεζικό ίδρυμα δανείζεται από τράπεζες με ενέχειρο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι κανόνες για τις εγγυήσεις που απαιτούνται. Οπότε το πώς θα αντιμετωπίσουμε εμείς με ένα συνολικό κανόνα είναι επίσης μια πρόκληση. Και ίσως με τη ρήτρα αυτή θα μπορούσαμε να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα ή να σκεφτούμε σοβαρότερα τα κουρέματα που ανέφερες ε, όταν υπάρχει δανεισμός έναντι μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή είναι η βασική τομή ε, στους οποίους θα μπορούσαμε να σκεφτουμε σοβαροτερα τα κουρεματα που ανεφερες οταν υπαρχει δανεισμος εναντι μετοχικου κεφαλαιου αυτη ειναι η βασικη τομη σε οποιους θα μπορουσαμε να συνεργαστουμε με τον Ρενάτο, αλλά νομίζω πως εργαζόμαστε για τον ίδιο σκοπό για την διαφάνεια δηλαδή και για να καταστεί ε, ο κανονισμός αυτός θετικός. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να μιλούν κάπως συντομότερα οι σκιώδεις γιατί θα πρέπει τώρα να έχουμε αρχίσει το επόμενο θέμα. Τέλος πάντων, ε, έχει τον λόγο η κυρία Σφίνμπορν. Είναι τεχνικό το θέμα. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχουμε. Έχουν πολλές λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάντως τον εισηγητή. Προσπάθησε να ισορροπήσει τα πράγματα. γιατί Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω ότι θα έπρεπε να έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε κάτι νωρίτερα. Έχουμε προσπαθήσει και στην προηγούμενη θητεία είχαμε διάφορα FSB, ERB και άλλες ευρωπαϊκές αρχές έχουν προσπαθήσει κάτι να κάνουν εδώ και μια εξαιτία από τα αιτία. Οπότε μέχρι τώρα έχουμε μια προσέγγιση αλλά χωρίς συνεργισμό. Έχουμε, είδατε τι έγινε με τα collaterals και είδαμε τι έγινε με τα ΡΕΠΟΣ για να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις αναφορές των συναλλαγών με τα FMD για τους ε, ε, επενδυτές. Οπότε ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα καλάθι και να μπορέσουμε να έχουμε τη σωστότερη ε, προσέγγιση. Συνόψιλον όλων αυτών, επομένως, να πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τους ορισμούς, γιατί έχουμε συζητήσει πολλά για το ότι θα πρέπει να αποδείξουμε ότι Όλα αυτά μπορεί να τα καλύψει η νομοθεσία. Είμαστε συνομοθέτες. Και θέλουμε να συμπράξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε τι είναι μία συναλλαγή για ομόλογα. Μην πάει στο επόμενο επίπεδο, το δεύτερο, ή το ξεκαθάρισμα του ορισμού. Επομένως, να μην σηκώσουμε τα χέρια και να αφαιθούμε στην σοφία της Κομισιόν και στην επόμενη φάση. Reduce ε, ε, ε, πώς θα γίνει η διάκριση μέχρι τώρα. Χρησιμοποιούνται εναλλάξ, αλλά έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Όμως έχουν τελείως διαφορετική νομική φύση. Άρα τουλάχιστον να συζητήσουμε για το κατά πόσον τελικά θα χρησιμοποιεί το reuse για να καλύψουμε και τις δύο έννοιες. Εάν θέλουμε να πάμε στην ορολογία του FSB, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε και τους δύο όρους, γιατί η κάθε έννοια έχει διαφορετική ρύθμιση. Άρα πάμε για δύο ορισμούς. Επίσης, αυτό που ανέφερε η Ντανούτα όσον αφορά την κοινοποίηση, γνωστοποίηση, πρώτα-πρώτα, προς την ρυθμιστική κανονιστική αρχή και δεύτερον προς τους επενδυτές. Να υπάρξει κάποια ρύθμιση και για τις δύο κοινοποίησεις γιατί όσον αφορά τα παράγωγα είχα μια αρνητική εμπειρία. Μόνο όταν ήρθαν οι δύσκολες ώρες κάναμε τη διάκριση τότε. Άρα θα πρέπει να υπάρξει σωστή ρύθμιση γιατί οτιδήποτε άλλο κοστίζει στους επαγγελματίες του κλάδου. Να υπάρχει με ένας ασφαλή δικαίου, να υπάρχει για τις ε, ρυθμιστικές αρχές κάποια σταθερότητα και άρα να χρησιμοποιήσουμε ό,τι ισχύει τώρα, αλλά το της κοινοποίησης θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Επίσης, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα διεθνή πρότυπα, όπως τους legal entry identifiers. Να, υπάρχουμε, έχουμε κάποιους κοινούς παρονομαστές παγκοσμίω. Επίσης και για το MIFID προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε το ότι εκεί θα υπάρξει στεγανή ρύθμιση και το ότι τώρα θα καλύψουμε περισσότερες συναλλαγές από ό,τι στην MIFID. Άλλο που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τους αντισυμβαλόμενους για χρηματιστηριακές και μη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Να δούμε τι ορισμό θα δώσουμε στον, στην έννοια του αντισυμβαλόμενου. Counterpart. αλλά να γίνει διάκριση και διασάφηση για να υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο. Επίσης, κάποια, κάποιες διατάξεις εδώ ισχύουν μόνο για τους συνελασσόμενους, για τους αντισυμβαλόμενους όσον αφορά χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αλλά υπάρχουν και άλλες διατάξεις που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες συναλλαγές. Για τις μη χρηματιστηριακές συναλλαγές θα πρέπει κάπως να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Να καλύψουμε και τις ΜΜΕ και αυτοί θα πρέπει να καλυφθούν. Άρα θα πρέπει και η έκθεση να μην επιβαρύνει τις ΜΜΕ υπερβολικά για αυτές τις προϋποθέσεις που θέτει. Για το κούρεμα, αναφέρεται εδώ πέρα το κούρεμα, haircut, κάτι το οποίο στην τελευταία διαβούλευση FSB συζητήθηκε. Μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, όμως τα κουρέματα δεν εμφανίζονται εδώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ε, θα θέλαμε. Οπότε τελικά, εάν εμφανιστούν στον κανονισμό ε, τα κουρέματα με αυτή την έννοια, τότε αυτό με ανησυχεί. Θέλουμε καλύτερο κανονισμό. Εάν θέλουμε να καλύψουμε ε, τα κουρέματα, τότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει το σχέδιο κειμένου, να το αντικαταστήσει, αφού κάνει αξιολόγηση των επιπτώσεων, με ένα άλλο κείμενο, το οποίο να καλύπτει τα κουρέματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αξιολόγηση επιπτώσεων. Crossover. Υπάρχει. Είναι πανταχού παρόν. Ως έννοια. Πανταχού παρούσα τέλος πάντων. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις προμήθειες της ΕΣΜΑ για κάποια καταπιστεύματα. Νομίζω ότι από την κερκόπορτα, από την πίσω πόρτα υπησύλθε αυτό στον κανονισμό. Δεν, είναι τόσο σωστό. Ίσως θα έπρεπε να πάει σε άλλη νομοθεσία για τα repositories. Επίσης, εάν έχουμε προμήθειες τέτοιες που να χρεώνονται, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός. Να μην υποκρύπτονται αυτές οι προμήθειες. Όπως κάνουν τώρα οι και αξιολόγησης. Είδαμε τι ρυθμίζεται μέσω του Μίφιλ για κάποιους ιδιωτικούς φορείς. Είναι πάρα πολύ τεχνικό το θέμα, πάρα πολλές ώρες θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε αυτά και περιμένω πώς και πώς να συνεργαστώ με τον εισηγητή. Ο την Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, διότι πολλά που είπαν η Ντανούτα και ο Ρενάτε με βρίσκουν σύμφωνο. Εδώ πρέπει να εντοπίσουμε τι ακριβώς θέλουμε να νομοθετήσουμε και να διευθετήσουμε. Δηλαδή, στην όλη συζήτηση για το συστημικό κίνδυνο, να σκεφτούμε πώς ακριβώς εντοπίζουμε τον ε, συστημικό κίνδυνο στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε σε πρώτη φάση σαφεί ορισμού, όχι μόνο στο επίπεδο 2, αλλά να είναι σαφέ το τι εννοούμε. Το είπε και, και οι ορισμοί που τώρα χρησιμοποιούμε πολλές φορές θα πρέπει να είναι απολύτως ελεγμένη και ε, βεβαιωμένοι και από νομική σκοπιά. Επίσης σημαντικό είναι εάν αυτός ο κανονισμός θέλουμε να ευθυγραμμίζεται με τους ισχύοντες κανόνες ε, να μην ξεχάσουμε το reporting και η υποχρέωση από πολλές εκθέσεων να είναι περιορισμένη για τους επενδυτές και τους παρόχους. Για τα κουρέματα νομίζω ότι έχει δίκιο η ΚΕΙ με την έννοια ότι αν το ζήτημα των κουρεμάτων το συζητήσουμε θα πρέπει να ε, υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο εδώ. Διότι έχω δει κάποιες προτάσεις που δεν συμπεριλαμβάνουν τα, ε, τα κρατικά ομόλογα προτιμησιακή μεταχείριση αυτών των ομολόγων όμως θα συνεχίσει να είναι ένα θέμα συζήτησης. Μπορούν να διακρίνονται από τα συνήθη χρηματοπιστωτικά προϊόντα, να εξαιρούνται από όλα και τα πάντα. Τα Υπουργεία και το Συμβούλιο ξέρω ότι επιθυμούν κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να γίνει μια επί συζήτηση και για τα κουρέματα. Επίσης κάτι άλλο που το έθιξαν και η Ντανούτα και η ΚΕΙ θα είναι βάση της συζήτησης είναι και το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, αν ε, θέλουμε νέε κατηγορίε, γραμμέ και νέε προτάσει εδώ, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν προτρέχουμε. Και να δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο, αλλά από τι μέχρι τώρα συνομιλίε μα θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, τη, τα χρονικά περιθώρια να τα σεβαστούμε και από τι δύο πλευρέ. Ε, Αυτέ ήταν οι δικέ μου παρατηρήσει για την ώρα και ε, μόνο για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε για την Γκουε Μαρίας Μαρίζα. Ευχαριστώ. Όχι, δεν θα λάβω εγώ το λόγο. Η συνάδελφό μου η Ειρήνα. Αλλά δυστυχώς είχε ένα προσωπικό κόλλημα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και ας συνεχίσουμε παρόλα αυτά διότι θα έρθει εκείνη σε επαφή με τον εισηγητή απευθείας. Πολύ καλά. Ε, τώρα να προχωρήσουμε λοιπόν στους πρασίνους η κυρία Ζολή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Καλωσορίζουμε την πρόταση ως ένα πρώτο βήμα στη βελτίωση της διαφάνειας ε, των δραστηριοτήτων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα αλλά να οδηγήσουν και σε σημαντικούς επικίνδυνους ε, συσχετισμούς μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των συνιστοσών τους που ανήκουν ε, στην σκιώδη τραπεζική δραστηριότητα. Είδαμε τα τελευταία χρόνια πώς ε, είναι απαραίτητη η καταγραφή πληροφοριών στα πλαίσια του, της προληπτικής εποπτείας όπως προβλέπει το SFT. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό σε συστημικό πλέον επίπεδο, να ληφθεί η σχετική πρόβλεψη και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και για όλους τους δρόντες σε αυτόν τον κλάδο. Κάποια ζητήματα πέραν της διαφάνειας τώρα, αναθεωρήσεις και καθεστώτα αφαιρεγιότητας για τα SFT, ειδικά εργαλεία SFT και δεσμευτικά εμ, δεσμευτεί κανόνες για την αξιολόγηση των εγγυήσεων και την διαχείρισή τους. Πιο συγκεκριμένα ως προς το πεδίο. Ίσως θα ήταν χρήσιμο το πεδίο αυτό να διευρυνθεί όπως είπαν πολλοί από τους σκιώδεις εισηγητές και στο πεδίο αυτό να συμπεριληφθεί η Κεντρική Τράπεζα, κυρίως για τους σκοπούς υποβολής εκθέσεων και την ε, ε, αποκάλυψη των συναθρισμάτων. Τώρα, για την SFT η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει τέτοιες οικονομικές προϋποθέσεις που να είναι ίδιες με τα κλασικά SFT, χωρίς ε, ε, παραθυράκια. Όμως χρειάζεται και καθοδήγηση επίπεδου 1 για να είμαστε σαφείς για το τι ακριβώς θα λαμβάνεται υπόψη μας προς τα κριτήρια. Η διαφάνεια προς τους επενδυτές είναι κάτι που ισχύει μόνο για τους επενδυτές στα κά και θα πρέπει να, να καλύψουμε εδώ όλους τους αντισυλα... αντισυμβαλωμένους σε αυτή ώστε να δημοσιοποιούνται ο όγκος, ο αριθμός, η ποιότητα και τα ε, στοιχεία που αποτελούν αυτούς τους τίτλους. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις ώστε οι αντισυμβαλόμενοι να δημοσιοποιούν σε συναθεσμένη μορφή την, ε, τα επίπεδα δανειοδότησης σε τίτλους όπως έδειξαν ότι χρειάζονται και τα τεστ κοπόσεως. Επίσης για τη διαφάνεια στα ρέπος θα πρέπει να προβλέψουμε τη δυνατότητα τέτοιας επαναγοράς τίτλων και να υπάρχει και συμμόρφωση με τις αρχές της ΕΣΜΑ και της EBCA. Ε, Η επαναγορά αυτή δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί την ε, ε, εμπορία της συναλλαγές για ίδιο λαγαριασμό. Ε, για την εποπτεία και τις σχετικές αρχές θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα άρθρο ώστε η να ζητά συνολικές εκθέσεις για τα ESFT ε για τον όγκο τους, για την αλληλοδιασύνδεση και τη σύνθεση των αντισυμβαλωμένων όπως προτείνει και το FSP Επιπλέον θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια διαφάνειας και να προσθέσουμε, να την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τα εξής. Εναρμόνιση, νόμοι αφαιρεγκαιότητα ως προς τα SFT ε, και καθεστώς super senior για κάποιες συνελλαγές ε, ρήπου καθώς και για, ποιότητα, για τις ποιότητας εγγύησης που προβλέπει η Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, αρχές εξυγίανσης στο ρήπο που αγοράζουν ε, ε, εγγύησης από τους ε, κατόχους των ρέπος πτωχευμένων ιδρυμάτων και τα ξαναπουλάνε επαναγοράζοντας έτσι το ενεργητικό των ιδρυμάτων που υποβάλλονται σε τεστ κοπόσεως. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη διαχείριση και εποπτεία και των εγγύσεων που παρέχουν τα διάφορα ιδρύματα. Σας αναπομονώ και εγώ για τη συμμετοχή μου σε αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστούμε και τώρα ο εισηγητής για την καταληκτή παρέμβασή του. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους που πήραν το για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. προφανώ ανυπομονώ και εγώ να συζητήσω τη συζήτηση μαζί του. Είδαμε ε, ότι παθιάζει και ενθουσιάζει πολύ τη συζήτηση αυτή, όπως και η προηγούμενη για τα διευθυντικά μέτρα για την βελτίωση τη ανθεκτικότητα των τραπεζών. Ακόμη βεβαίω και αν είναι πολύ διαφορετικέ οι απόψει. Προσπαθώ να δω την όλη συζήτηση όχι απλώ ω ένα τεχνοκρατικό ε, σημείο με κάποιε πτυχέ που κάποιε φορέ είναι και κατανόητε όσου ε, στον επαγγελματικό του βίου δεν έχει υπάρξει οικονομολόγο. Θα ήθελα τη συζήτηση αυτή να τη βλέπω σε ένα μέρο αυτή τη ε, διαπίστωση που μα υπενθύμησε το πρωί ο, Χόκ, ο κ. Χόκμαρκ. 800 δι λείπουν από τι επενδύσει για την πραγματική οικονομία. 800 δι λοιπόν στι επενδύσει για τη δημιουργία θέσει απασχόληση, για τον πλούτο και την ευημερία που τόση ανάγκη έχουν όλοι οι λαοί τη Ευρώπη. Αυτό δεν θα συμβεί εάν δεν υπάρξει εμπιστοσύνη την οποία όλοι ζητήσαμε για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για του επενδυτέ τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια και για όσα Πιστεύω ότι θα πρέπει να εκπροσωπεί το τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή δημιουργία πλούτου και θέσεις εργασίας, όχι αυτοεξυπηρέτηση. Τα αυτήν την ε, οπτική γωνία νομίζω ότι μπορούμε να δούμε την όλη μας συζήτηση και τα στοιχεία της που φαίνονται απλώς τεχνοκρατικές λεπτομέρειες αλλά στην πραγματικότητα αυτό το νομοθέτημα βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματο. Δημιουργία ευημερία, δημιουργία πλούτου, με δημιουργία θέσει απασχολήσει που λείπουν στην Ευρώπη. Πρέπει να αναθερμαθούν οι επενδύσει με μεγαλύτερη ε, στήριξη τη εμπιστοσύνη, τη αμοιβαία εμπιστοσύνη που λείπει μεταξύ των πολιτικών ηθινόντων, αλλά και μεταξύ χωρών όπω φαίνεται. Μεταξύ των ε, ε, παραγόντων του τραπεζικού κλάδου, μεταξύ των επιμέρου ε, μερών. Ε, λύπη μεταξύ τραπεζών και επιχειρήσεων. Ε, υπενθυμίστηκε το πρωί και μας είπε ο πρόεδρος του London Stock Exchange ότι υπάρχει ένα σωρό χρήμα για την αγορά. Γιατί όμως οι τράπεζες δεν έχουν εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις και δεν δανείζουν. Οι επιχειρήσεις ε, μπορούν πολλές φορές να δανειστούν χρήμα αλλιώ από την αγορά ενδεχομένω, αλλά αν δεν τι έχουν εμπιστοσύνη να αναβάλουν τι επενδύσει. Ένα φαύλο κύκλο λοιπόν, ο οποίο πρέπει να έρθει. Αυτό το νομοθέτημα δεν είναι απλώ ένα τεχνοκρατικό στοιχείο, αλλά και μια προσπάθεια να οδηγηθούμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης αυτής είναι το ίδιο με την προηγούμενη. 21 Ιανουαρίου σχέδιο, 27 προθεσμοί για τροπολογίες, 23 Φεβρουαρίου εξέταση τροπολογιών, 23 Μαρτίου ψηφοφορία και στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Τώρα περνάμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πάρα πολύ σημαντικό. Έκθεση για την εξέταση του πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης ε, απολογισμός και μελλοντικέ προκλήσεις. Όπως ξέρετε, εξετάζοντας το εξαπλό πακέτο, η Κομισιόν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα του νομικού πλαισίου και την πρόοδο για τον στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και η Επιτροπή μας αποφάσισε να συνεισφέρει ε, και βεβαίως αυτό να γίνει εγκαίρος με μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Ε, Ευχαριστώ που βάλατε το θέμα αυτό για πρώτη ε, ανταλλαγή απόψεων στη μέση διάταξη. Αυτό το οποίο θέλουμε όταν ε, καταλήξαμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα ήταν το ότι θέλαμε και εμεί να κινηθούμε στα πλαίσια αυτή τη δυναμική για το κείμενο εκείνο το οποίο είχαμε ξεκινήσει στην προηγούμενη ε, θητεία για να έχουμε κάποιε συναντήσει και γι' αυτό στις 14 του είχε την αξιολόγηση η Κομισιόν του για το, για το πρώτο ή το δεύτερο πακέτο εξαπλώ των μέτρων, το six pack και επίσης ε, ε, έχουμε συνεργαστεί με συνάδελφους και σκιώδης πριν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορέσει να μας υποβάλει αυτή την πρώτη αξιολόγηση όσον αφορά τα μέτρα τα οποία εμείς έχουμε εγκρίνει οπότε γι' αυτό και παρουσιάσαμε ένα πρώτο εγγραφό εργασία. έτσι έχουμε εδώ πέρα δεδομένο το, το, το πλαίσιο της προβληματικής για να δούμε πού θα δουλέψουμε για να δούμε τι θα γίνει με τα επιμέρους θέματα. Γιατί τελικά έτσι θα πρέπει να δουλεύουμε με τα έγγραφα εργασία, γιατί αυτό θέλαμε να κάνουμε, να είμαστε ειλικρινεί και αποφασιστικοί όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ότι ε, τα ξέρουμε εμείς εδώ στην Οικονομική Νομιστική Επιτροπή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει τη μακροοικονομική κρίση, δεν είχε τα, προσόντα ούτως είπε, τα εργαλεία στην προηγούμενη θητεία. Οπότε αυτό το οποίο τώρα τίθεται σαν ερώτημα είναι πώς αξιολογούμε ε, ε, της, ε, την ομοθεσία την οποία έχουμε θεσπίσει και σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας του 2005 και κατόπιν με το 6 Pack, το 2 Pack ε, όσον αφορά επίσης τη, τόσο έχουμε θεσπίσει το δημοσιονομικό είπαμε επομένως ότι θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το μείγμα πολιτικής το οποίο τώρα αναδύεται με όλα αυτά οπότε παρακαλώ εξετάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο του Οκτωβρίου 2013 της Επιτροπής εκεί ε, έχει εύστοχες παρατηρήσεις όσον αφορά όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στην Ευρωζώνη. Οπότε τα ζήματα που έχουν να δούμε είναι κατά πόσον τώρα με αυτό το πλαίσιο μπορούμε να έχουμε το καλύτερο μείγμα πολιτικής. Εάν έχουμε κάτι για τα δικυκλικά φαινόμενα, εάν επίσης υπάρχει το επίπεδο το οποίο χρειάζεται, ώστε οι χώρες οι και οι να προσαρμοστούν. Οπότε γι' αυτό και κανονίσαμε ε, αυτό το χρονοδιάγραμμα, ε, αυτού του συνάντηση που είναι τριπλή. Πρώτα-πρώτα έχουμε αυτές τις, τις επίσημες συναντήσεις σε σχέση με τα κείμενα για την εξαπλή δέσμη, τη διπλή δέσμη, να υποβάλει την προτασίδηση η Επιτροπή όχι μόνο για την αξιολόγηση του τι έχει γίνει, αλλά για να ε, προταθούν και για να θεωρούν ε, κανονισμών, ακριβώς όπως ο ίδιος ο κανονισμός επιτάσσει. Επίσης, δεύτερη διάσταση είναι ε, τι αποφάσισε τον Ιούνιο το Συμβούλιο. Μας πρότεινε να δούμε τι περιθώριο ευελιξίας υπάρχει σήμερα. Επίσης, τρίτη πτυχή είναι αυτό το οποίο αποφάσισαν οι συντονιστές αποφάσιζαν για αυτόν τον τίτλο της έκθεσης, για μια γενικότερη, ευρύτερη προσέγγιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ τους συντονιτές μας γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ε, έναν πρώτο προβληματισμό. Θα επανέλθω σε αυτό. Οπότε, με αυτή την προσέγγιση θα πρέπει επίσης να καλύψουμε κάποιες προτάσεις που έχουν από άλλες πλευρές προταθεί και επίσης το δούνου του, το οποίο συμφωνεί ότι το, τις δημοσιονομικές επιπτώσεις και τα απολογιστικά αποτέλεσματα κάποιων μέτρων δεν τα εκτιμήσαμε σωστά. Επίσης, λάβουμε υπόψη τι είπε ο πρόεδρος της ε, Κεντρικής Τράπεζας τότε στο Τζάκσον. Ε, τι είχε πει τον Αύγουστο ο πρόεδρος εκτός Ευρώπης το είπε. Euh, για το ότι δεν ελήφθη αρκετά υπόψη η μεταβλητή της συνολικής ζήτησης. Οπότε να δούμε επομένω στο σύνολό του το θέμα αυτό το οποίο έχουμε με τις τραπέζες και να δούμε τι προτάσεις έχουμε αλλά και τι εργαλεία μέσα πολιτικής έχουμε. Υπάρχει ε, υπάρχουν κάποια μέτρα προληπτικού χαρακτήρα του συμφώνου. Έχουν την αναγκαία ευελιξία ή οφείλουμε να τους την προσδώσουμε εμείς. Επίσης, Κατόπιν των διαπραγματεύσεων, όταν εγκλέμε το την εξαπλή και την διπλή δέσμη, στη συνέχεια είχαμε την επιστολή Ρεν. Ενδιαφέρον γιατί τώρα είναι συνάδελφος εδώ στο Κοινοβούλιο. Για να μας κάνει αυτός μια αυθεντική ερμηνεία λοιπόν σε αυτήν την ε, επιστολή σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς είπαμε για τις επενδύσεις. Από τότε γίνανε πολλά. Και τότε εμείς φοβόμασταν ότι οι φόβοι μας θα υλοποιηθούν. Είχαμε αυτού του είδους την ρήτρα επένδυσης της επιστολής Ρεν. Όμως αλλάξαν τα πράγματα. Άρα για να δούμε. Μήπως για τις επενδύσεις ήταν υπερβολικές οι τότε απαιτήσει. Άρα, για να δούμε τι θα γίνει με το περιθώριο λιγμών που έχουμε, τι θα πει η εξαιρετική υπερίσταση, unexpected adverse economy event, απροσδόκητο οικονομικό φαινόμενο, πώς ορίζεται αυτό, όλες αυτές τις διάφορες μεταβλητές για να λάβουμε υπόψη επομένως ότι θα γίνει για τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επιπτώσεις που είχαν οπότε έγιναν επί των οικονομιών. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τα προληπτικού χαρακτήρα δημοσιονομικά μέτρα. Γιατί θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση όσον αφορά την δράση που ανέλαβαν τα κράτη-μέλη για να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, άλλη προβληματική είναι η οικονομική πραγματικότητα που σήμερα μας περιβάλλει. Πρώτα-πρώτα, με υψηλός πληθωρισμός, χαμηλή ανάπτυξη και χαμηλή απασχόληση. Το χρέος Τι είναι, είναι συνέπεια του χαμηλού πληθωρισμού, τι γίνεται. Γιατί μιλούμε για πολλά θέματα, πολλά ερωτήματα που αναδύονται και θα πρέπει να απαντηθούν. Ε, νομίζω ότι μακρηγόρησα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι λένε και οι πανεπιστημιακοί, γιατί και αυτοί έχουν υποβάλει πολλές προτάσεις όσον αφορά το πού θα πρέπει να προτεραιότητα ούτως ώστε να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε για την οικονομική διακυβέρνηση. Ορισμένοι προβληματίζονται για το τι θα πει πίθε εν δυνάμει ανάπτυξη το κατά πόσον έχουμε κάποιο είδου ε, αυτόματη αναδιάρθρωση του χρέους. Άλλοι λένε για μια νέα προσέγγιση στα πλαίσια του ισχύντος νομοθετικού πλαισίου, ούτως ώστε να έχουμε άμεση μείωση των φόρων και βαθμία μείωση των δαπανών, αλλά έτσι θα έχουμε την... θα πρέπει να έχουμε μία παρέκκληση από την, χαρα... από την επιβαλλόμενη πολιτική. Το λένε αυτό λοιπόν πανεπιστημιακοί κύκλοι και ότι τελικά τα κράτη που έχουν μισονομικό περιθώριο θα πρέπει να κάνουν επενδύσεις, κρατικές επενδύσεις, ούτω ώστε κυρίως να μπορέσουν να μειώσουν αυτό που μας έχει πλήξει, δηλαδή την έλλειψη επενδύσεων. Είναι κατακλείδη. Πρόεδρε, έχουμε την τρίτη διάσταση της έκθεσης. Έχουμε τις σχετικές διαπιστώσεις, είπαμε για την προβληματική για την ευελιξία, αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα πούμε ως Επιτροπή για την διακυβέρνηση. Την οικονομική διακυβέρνηση είμαστε στην αρχή της θητείας. Δεν είπα ότι θα πρέπει να ανοίξει το κτίριο της Πανδώρας, αλλά μια που είναι αρχή της θητείας θα πρέπει να τεθούν επιτραπέζεις κάποια βασικά ζητήματα. Έχουμε την ανακοίνωση του 2012 για το blueprint έκθεση Tyson. Ακόμα δεν κατέληξαν πουθενά όλες αυτές οι πρωτοβουλίες. Άρα θα πρέπει να είμαστε εύστοχοι στις αναλύσεις μας για να κάνουμε κάτι παραπάνω από ένα βραχυχρόνιο μέτρο για να μην ξαναβρεθεί μπροστά σε διέξοδο μεσοπρόθεσμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα-πρώτα να έχουμε νέα εκτροπή των δημοσιονομικών, ε, επίσης να έχουμε και πάλι μια ανυπόφορη ε, απόκληση των κρατών μελών για τα δημοσιονομικά και τρίτον να έχουμε αυτή την, την χρόνια έλλειψη ε, επενδύσεων. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Και τώρα ο λόγος στον πρώτο μιλητή, η κυρία Ντελάγκε, η συγκεκριά του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγητρία για αυτό το έγγραφο εργασίας που το βρίσκω μια πολύ καλή βάση για τη συζήτησή μας. Την έκθεση την περιμένουμε, όπως είπαμε, το Δεκέμβριο. Στρέφουμε λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελπίζοντας όντως το Δεκέμβριο να την ε, δημοσιεύσει για να ακολουθήσει και η δική μας έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η Νομισματική Ένωση ήταν περισσότερο νομισματική παρά δημοσιονομική, ούτε και καν οικονομική φυσικά κατά τη στιγμή της δημιουργίας της να σας πω και μια ιστορία από την προσωπική μου εμπειρία. Ξέρω την ευαισθησία και των 100 μελών για τα θέματα αυτά. Εγώ τότε με σπούδαζα σε ασπό το 1995 στη Γαλλία και μια από τις τελευταίες μου πτυχιακές, ο τίτλος είχε τίτλο μάλλον, ε, ε, ζητήθηκε να έχει από τον καθηγητή μου, θα πρέπει να στραφεί προς την νομισματική προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε ε, η συζήτηση αυτή ότι δεν θα είχε καν ε, ξεκινήσει σε ένα Ολλανδικό πανεπιστήμιο, έτσι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι κάποιοι κανόνες υπήρχαν στην αρχή της νομισματικής ένωσης, όπως για το δημόσιο χρέος, τα δημόσια ελλείμματα, τα κρατικά ελλείμματα. Δεν ε, συμφωνούσαν και συμπορθώνονταν βεβαίω με όλα αυτά τα, όλα τα κράτη-μέλη, στα μέσα της περασμένης δεκαετίας εννοώ. Γι' αυτό και προέκυψαν κάποια τα προβλήματα που είδαμε στη συνέχεια. Αυτό επίσης δείχνει την σαφή σχέση μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών σε αυτό τον τομέα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Τα κράτη-μέλη, και είναι σαφής μου πεποίθηση αυτή, δεν μπορούν να ε, μετατοπίζουν τις ευθύνες τους σε στοιχεία που οι ίδιοι δεν μπορούν να επιλύσουν ε, σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην επιτρέψουμε να χρησιμοποιούμαστε ε, να γινόμαστε αντικείμενα εκμετάλλευση. Σε αυτά τα δύο επίπεδα, το εθνικό και το ευρωπαϊκό, θα πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία. Μόνο τότε υπάρχει η δυνατότητα να ενισχύσουμε τι οικονομίε μα. Νομίζω ότι το εθνικό στοιχείο είναι ένα από αυτά που πρέπει να ε, καλυφθεί λίγο περισσότερο στην έκθεση. Επίσης να μην ξεχνάμε γιατί το τωρινό σύστημα της οικονομικής διακυβέρνησης δημιουργήθηκε. Το Six και το Two δημιουργήθηκαν αφού πολλά κράτη-μέλη σχεδόν ε, πτώκευσαν λόγω του χρέους τους ή τέλος πάντων απέκλειναν των στόχων του χρέους. Ε, αυτό οδήγησε σε καταστροφή στα συγκεκριμένα κράτη-μέλη αλλά ε, και σε κλειδονισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο. Τα κράτη-μέλη αυτά ξέφυγαν ε, χάρη στη δημιουργία των μηχανισμών σταθεροποίηση όπω τον ESM. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι το Τούπα και το SIXPAC στο σκοπό είχαν να αποφύγουμε την επανάληψη τέτοιων εξελίξεων. Σαφώ είναι σημαντική η δημοσιονομική πειθαρχία. Έπρεπε να ενισχυθεί, αλλά και άλλοι παράγοντε πρέπει να ληφθούν υπόψη όπω οι μακροοικονομικέ ανισορροπίε. Οι ανισορροπίε αυτέ όμω μετρώνται εντό χωρών και όχι συγκριτικά μεταξύ χωρών. Μην ξεχνούμε ότι πραγματικά αίτια της κρίσης ήταν η μη, τα μη βιώσιμα κρατικά δημοσιονομικά και οι μη βιώσιμες ε, ανισορροπίες ε, στις και αποκλήσεις μεταξύ των κατομελών. Αυτό να το λέμε και μάλιστα δυνατά. Τέτοιες μακροοικονομικές λοιπόν ε, ε, αποκλήσεις πρέπει να συνοδεύονται από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Όχι γιατί δεν μας αρέσουν οι κρατικές δαπάνες, οι κρατικές δαπάνες βεβαίω πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο, ε, αλλά αυτό είναι κόκκινη γραμμή για μας. Πρέπει να προσέξουμε και να μην επιβαρύνουμε τις επόμενες γενιές με επίπεδα χρέους που δεν μπορούν να αντέξουν. Νομίζω, και εδώ στρέφομαι σε αυτά που νομίζω θα πρέπει να μας απασχολήσουν κατά κύριο λόγο στην έκθεση, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας που αξιολογούμε την αποτελεσματικότητά της για να αποφύγουμε στο μέλλον οποιαδήποτε κατάσταση απόκλησης ως προς το χρέος για μια χώρα. Δηλαδή να αξιολογήσουμε σωστά τα πορίσματα του Τούπα και του ΣΥΚΣΠΑΚ, κάτι που ήταν και πραγματική ε, αποστολή της ρήτρας αναθεώρησης. Έγιναν κάποιες χώρες κάπως πιο ανθεκτικές ή ακόμη κινδυνεύουν να πτωχεύσουν λόγω του χρέους τους. Τα ελλείμματα κατέβηκαν κάτω από την πρώτο του 6%, τα το 60% και τα κράτη με τις χώρας συστάσεις συμμορφώνονται ή όχι, ιδίω προς τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Εγώ προερχόμαι από ένα μικρό κράτος μέλος. Πρέπει να πω ότι σημαντικό είναι και οι μικρές με τις μεγάλες χώρες να έχουν την ίδια μεταχείριση. Και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά ε, υλοποιεί τους κανονισμούς και το κάνει και στο μέλλον. Δεν είναι βεβαίως αυτός ο οριστικός τελικός κατάλογος, αλλά είναι μια σειρά από ερωτήματα που θα θέλαμε να καλύπτονται. Βεβαίως είναι νωρίς για να αξιολογήσουμε κάτι που μόλις δύο χρόνια λειτουργεί, αλλά και πάλι ευχαριστούμε πολύ για την διεξοδική σας δουλειά, για τα έγγραφα εργασίας. Ε, ανυπομονώ για τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερως για τις απόψεις των συναδέλφων. Όπως ε, είπα δυστυχώς ε, για τους υπόλοιπους που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση πρέπει να πω να υποδεχτώ έναν υπουργό στις 12 αλλά οι συνεργατές μου θα παραμείνουν και με τα χαράς να συζητήσω με οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να έχουμε συνομιλίες για το ζήτημα αυτό εκτός της συγκεκριμένη συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και όλους τους υπολείπους που συμμετέχουν. Thank you. Now the next speaker, Mr. Ευχαριστώ, Bernd για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύρια Μπερές για την έκθεση αυτή. Σωστά είπατε πως είναι μια έκθεση που ανοίγει μια συζήτηση στην οποία θα ήθελα να συνεισφέρω και εγώ. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε πως η έκθεσή σας βάζει κάποια πράγματα, δηλαδή μιλάτε για την έλλειψη ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και μετά συνδέεται ε, το θέμα αυτό με τις αιτίε. Η απάντησή σας έρχεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι το θέμα του αποτελεσματικότερου μείγματος πολιτικής ε, και λέτε πως εντός της Ευρωζώνης θα πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσματικότερο μείγμα πολιτικής, ε, ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, δεν είναι το κατάλληλο και ειδικά στον τομέα τον δημοσιονομικό πρέπει να υπάρξει μια πιο επεκτατική πολιτική και μετά λέτε να εκμεταλλευτούμε την ευελιξία που υπάρχει στα 2 pac και λοιπά μια σειρά προτάσεων και είναι θετικό. Μα, μα κάνετε μια σειρά προτάσεων και λέτε με ποια κριτήρια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία και λέτε πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους ορισμούς και το ότι δεν υπάρχει αρκετή ακρίβεια και να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να δικαιολογήσουμε μια πιο επεκτατική πολιτική, δηλαδή ακόμα περισσότερα χρέη. Καλό είναι, νομίζω, πως ε, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις εδώ. Και το νόημα βεβαίως δεν είναι να ψάχνουμε συνεχώς πόσο περισσότερο μπορούμε να χρεωθούμε με βάση τους υφιστάμενους κανόνες, αλλά να δούμε και ποια ήταν η πρόθεση του νομοθέτη όταν εγκρίθηκε το διπλό και το εξαπλό πακέτο και πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ακριβείς τους όρους και τις διατάξεις για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόθεση. Και βεβαίως μετά στο επόμενο μέρος της ε, έκθεσης μιλάτε για δημοκρατική λογοδοσία και αυτό πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Και να σας πω τι λείπει κατά την απόψή μου από την έκθεση αυτή. Μιλάτε για την έλλειψη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και εδώ πέρα υπονοείται βεβαίως πως η Ευρωζώνη αναπτύσσεται αργότερα από άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στις περιοχές εκείνες που έχουν καλύτερη ανάπτυξη εντός της Ευρωζώνης. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη εκείνα που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη και να δούμε τι ανάπτυξη περιέχουν και βέβαια μετά να δούμε πού οφείλεται η διαφορετική ανάπτυξη. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή μεταξύ αυτών που είναι εντός και εκτός της Ευρωζώνης και πού οφείλεται αυτό. Και ερχόμαστε έτσι στο ερώτημα του εάν είναι το ενδεδειγμένο το μείγμα της πολιτικής που έχουμε στην Ευρωζώνη. και βεβαίως μπορούμε να δούμε τα νομισματικά και τα δημοσιονομικά μέσα που έχουμε στην ζώνη μας. Βλέπουμε λοιπόν πως τα κράτη εκτός Ευρωζώνης ακολουθούν λιγότερο επεκτατική νομισματική πολιτική από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Οπότε τίθεται το ερώτημα Πού οφείλεται το ότι εκτός της Ευρωζώνης είναι καλύτερη και ευνοϊκότερη η ανάπτυξη από ό,τι εντός. Και τίθε το ερώτημα του εάν έχετε δίκιο ε, σε αυτό που λέτε πως δεν έχουμε ανάπτυξη λόγω του μείγματος της πολιτικής. Εγώ θεωρώ λοιπόν πως θα πρέπει να μιλήσουμε για άλλες αιτίες ε, που θα εξηγήσουν την έλλειψη της ανάπτυξης να δούμε ποια θα είναι τα κίνητρα που απαιτούνται για να υπάρξουν επενδύσεις, ε, γιατί συνεχώς λέμε πως δεν υπάρχουν επενδύσεις. Πρέπει να μιλήσουμε για την υπερβολική φορολόγηση, τις υποδομές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά στην Ευρωζώνη, να μιλήσουμε για την έρευνα και την ανάπτυξη, για τα κίνητρα που ε, οδηγούν σε ανησυχητική χρέωση των ιδιωτών και βέβαια αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Φον Βαστσέκερ, δηλαδή την κρίση εμπιστοσύνης στα χρηματοπιστωτικά μας ιδρύματα και ειδικά τις επενδυτικές τράπεζες. Όλα αυτά είναι εμπόδια για να επιτύχουμε ε, ιδιωτικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για το μοναδιαίο κόστος εργασίας και τι επίδραση έχει στην διεθνή ανταγωνιστικότητα. Μιλήσατε για μια επανισορρόπηση για να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και είπατε πως θα πρέπει να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και τα πιο ανταγωνιστικά κράτη-μέλη θα πρέπει να τονίσουν την εγχώρια ζήτηση. Το να τονώσουμε την εγχώρια ζήτηση βεβαίως δεν είναι παρά ένας εφημισμός ε, για κρατικά μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν ψηλότερα το επίπεδο των τιμών. Τι σημαίνει αυτό στο διεθνές ε, πλαίσιο. και πώς θα επιδρούσε αυτό στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των κρατών μέλων. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχει μεγάλη σημασία αυτό το ζήτημα, γιατί η πολιτική δημοσιονομική είναι μία μέθοδος για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές ανταγωνιστικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι σημαντική και πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Και βέβαια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η πρόταση λοιπόν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ασκήσει τέτοια πολιτική είναι μια ιδέα η οποία δεν συμβιβάζεται με την κατανομή των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βεβαίως εδώ πέρα έχουμε μια α, σαφή υπεροχή της αρχής της επικουρικότητας. Θα ήθελα να πω πως ο πολλαπλασιαστής ε, ο λεγόμενος ε, των κρατικών δαπατών, δαπανών δεν είναι κάτι το μηχανικό που δρά αυτομάτως εξαρτάται οπωσδήποτε από την οικονομική συγκυρία και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και βεβαίως υπάρχει σαφής διαφορά στην επίδρασή του ανάλογα με την φάση του οικονομικού κύκλου στην οποία βρισκόμαστε. Οπότε δεν είναι καθόλου βέβαιο πως μια τέτοια πολιτική θα έχει ακριβώς ε, την επίδραση την οποία θέλετε. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ Έχουμε επίσης ε, το ζήτημα της ε, ευελιξίας στο οποίο είσαστε πράγματι ε, υπέρ. Βεβαίως η πρόθεση εδώ πέρα ήταν του νομοθέτη να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του χρέους. γιατί μην ξεχνάμε πως περισσότερα χρέη σήμερα σημαίνει περισσότερα τοκοχρεολύσια αύριο. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η δυναμική του χρέους η οποία μπορεί βεβαίως να μας οδηγήσει σε, στον πειρασμό του να έχουμε χαμηλότερο χρέος ή αντιθέτως να χρεωθούν περισσότερο σήμερα επειδή είναι χαμηλά τα επιτόκια αλλά να βρεθούμε αύριο αντιμέτωποι με πολύ υψηλότερα επιτόκια και να οδηγηθούμε εκ νέου σε όξυνση της ε, κρίσης. Ε, τέλος, να έρθω πράγματι στο θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας. Εδώ πέρα συμφωνώ πλήρως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ειδικά η Κομισιόν, να δίνουν λογαριασμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις επιτροπές του. Και ακριβώ εδώ πέρα πρέπει να ε, παρουσιάζονται σαφώς τα γεγονότα. Και θα ήθελα εδώ πέρα να πω το εξής για τις συζητήσεις που θα γίνουν με την Κομισιόν τον Δεκέμβριο. Πρέπει να παρουσιαστούν απλά τα δεδομένα. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων είναι κάτι το διαφορετικό και θα πρέπει να γίνει μια κριτική ανάλυση. Ε, τώρα για συμπέρασμα βέβαια δεν θα επαρκεί ο χρόνος και οπωσδήποτε χρειάζεται και λογοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων στα δικά τους κοινοβούλια για να προκύψει σαφώς το ποια μέτρα θα ληφθούν, με ποια κίνητρα λαμβάνονται και τι θα προκύψει ως συνέπεια για την ανταγωνιστικότητα των εν κρατών, για το φορολογικό βάρος, καθώς αυτά χρηματοδοτούνται από φόρους και βέβαιω για τις μελλοντικέ γενναίες που θα φορτωθούν το χρέος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Τόιρε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Μπερές και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος των φιλελευθέρων για την δουλειά που έχετε κάνει. Θα ήθελα να πω πως μία νομισματική ένωση βεβαίως μπορεί να δημιουργήσει και, και πρέπει να δημιουργήσει και μια πολιτική ένωση. Γι' αυτό ακριβώς η νομισματική μας ένωση ε, απέτυχε γιατί υπήρχε μια υπανάπτυξη των αντίστοιχων πολιτικών θεσμών. Και βεβαίως Όλα αυτά ξεκίνησαν το 2013 με τη Γαλλία και τη Γερμανία που παραβίασαν τις συνθήκες και δεν εμποδίστηκαν. Αυτή ήταν η αφετηρία της αυστηροποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και η οποία μετά μεταφράστηκε σε νομοθεσία. Βεβαίως ε, το χρόνος ο οποίος πέρασε είναι πάρα πολύ λίγος για να κάνουμε μια πραγματική αξιολόγηση της νομοθεσίας. Οπότε και εμείς συμφωνούμε με την κυρία Εστέρ Ντελάνγκε πως πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και βεβαίως είδαμε πάρα πολύ εντατικά αυτές τις στάσεις αναχώρα και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι πώς θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Εδώ πέρα παραδείγματος χάρη η Κομισιόν mm. είπε για τη χώρα μου, τη Γερμανία, πώς οι επενδύσεις είναι χαμηλότερες από τις ε, αποσβέσεις, οπότε ε, ουσιαστικά δεν κάνουμε αρκετές επενδύσεις και το ερώτημα είναι ακριβώς πώς ε, μπορούμε να δώσουμε μια όθηση στις επενδύσεις, κάτι το οποίο δεν συζητιέται αρκετά στην χώρα μου. και βεβαίως είχαμε ακριβώς αυτή την μείωση του φορολογικού κόστους προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες και αν δεν εφαρμόζονται το γιατί όχι. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει μια συνολική αμφισβήτηση του πλαισίου ή αν χρειάζεται μια χαλαρωσή του. Εμείς διαφωνούμε και με τα δύο αυτά πράγματα τα οποία λέτε. Εμείς θεωρούμε πως είναι η καλύτερη πολιτική αυτή για το μέλλον. Και βεβαίως ε, πρέπει να συζητήσουμε για τον ρόλο των ε, κεντρικών ε, τραπεζών και να δούμε αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Λούκε, δηλαδή γιατί αναπτύσσονται οι χώρες εκτός Ευρωζώνης. Εγώ σκέφτομαι αμέσως την Ευρωζώνη που έχει σαφώς χαλαρότερη νομισματική πολιτική με την ποσοτική χαλάρωση. Μιλάμε για 250 δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες. Αν υπολογίζαμε το ίδιο στην Ευρωζώνη θα μιλούσαμε για αγορά κρατικών ομολόγων για πάνω από ένα 1,43 εκατομμύρια ευρώ, κατά το οποίο δεν έγινε. Και νομίζουμε πως ούτως ή άλλως έτσι θα ξεπερνούσε την εντολή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πρέπει άρα να δούμε ποια θα είναι η μελλοντική της εντολή. Κατά την άποψή μου η αποστολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιμών. Δεν είναι αποστολή της να χρηματοδοτεί χώρες και δεν είναι η αποστολή της η πολιτική απασχόλησης. Έτσι δεν είναι η ίδια αποστολή με το Αμερικάνικο Fed. Όσον αφορά τις ε, δημόσιες επενδύσεις και το κατά πόσο μπορούν να κινητοποιήσουν την οικονομία, πρέπει να δούμε ακριβώς το εάν έχουν αυτή την επίδραση και αν ναι, πώς μπορεί ακριβώς να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνητρο, αν θα είναι δηλαδή μια αποκοπήν αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, κάτι για το οποίο δεν είμαστε υπέρ. Εμείς θεωρούμε πως αυτή η πολιτική έχει φτάσει στα όρια της. Ίσως στρατηγικά σε κάποια σημεία, συνέρευμα και ανάπτυξη και στις υποδομές να μπορούσαμε να το κάνουμε επίσης. Θα πρέπει να μας ανησυχήσει πως ε, οι πολίτες ε, κάποιων ε, χωρών ε, πλήρωσαν ε, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη Σλοβακία, στη Λιθουανία, στην Ισλανδία τακτοποίησαν τα οικονομικά τους ε, και δεν νομίζω πως είναι σωστό να πληρώνουν για άλλες χώρες που δυσκολεύονται να αναλάβουν ανάλογες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω έτσι άρα πως μπορούμε να έχουμε μία βάση ε, για μία πολιτική τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Σύμφωνο Το Τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω αφορά τις κρατικές χρεοκοπίες. Ε, πράγματι κάποια κράτη-μέλη εξακολουθούν να έχουν πάρα πολύ υψηλό και ανισχυτικό χρέος ε, ακόμα και σε κάποιες χώρες που φαινομενικά είναι στιβαρές οικονομικά όπως η Γερμανία είναι ανησυχητικό το ζήτημα και θα έπρεπε ίσως να δούμε τι μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις χρεοκοπίας κρατών εμείς θεωρούμε πως δεν έχουν γίνει εδώ πέρα αρκετά πράγματα για να Ε, έχουν και οι ιδιώτες πίστοτες. Θα τα δούμε αυτά και με τους κοιόδης εισηγητές και θα κάνουμε τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η ε, κυρία Ματίας για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας την εισηγήτρια για την πρόταση που μας έχει υποβάλει. Νομίζω ότι μία ότι η πρόταση είναι καλή και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διάρθρωση και τα ζητήματα που γύρει. Γι' αυτό θα ήθελα να σχολιάσω κάποια από τα ζητήματα που αναφέρονται στο έγγραφο. Αλλά και κάποια από αυτά που ανέφεραν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Όταν συζητούν το κατά πόσο είναι εύστοχο ή όχι, να γίνει οποιαδήποτε αναθεώρηση ή αξιολόγηση του όλου πακέτου τη όλη δεσμή μέτρων για την οικονομική διακυβέρνηση. Όχι απλώ είναι εύστοχο, είναι υποχρεωσή μα να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει ε, να δούμε και κάποια από αυτά που αναφέρει η έκθεση, η συγκήτρια στην ε, εισαγωγή, στο προήμιο κάνει κάποια γενικά σχόλια για το τι συνέβη μετά το Μάστριχτ, τις δυσκολίες ε, ανάπτυξης, τις ε, δυσκολίε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και της ε, ρήτρα bailout, ώστε τα δημοσιονομικά προβλήματα ενό κράτου της Ευρωζώνη να μην έχουν επιπτώσεις στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή να μην υπάρχει μετάδοση των προβλημάτων. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάποια χρόνια μετά και στην οικονομική κρίση είδαμε να γίνεται το αντίθετο. Όχι απλώς ε, υπήρξε μετάδοση, αλλά ήταν και συστηματική και αυτόματη αυτή. Ήδη, ε, μόλις πέρσι, μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το νομοθετικό πακέτο ήρθε χωρίς να υπάρχει ένα σύνολο στόχων, συγκεκριμένων σκοπών οι χώρες σε πρόγραμμα με τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να επιφέρουν, με διευθυντικές μεταρρυθμίσεις, πολλές από αυτές ξεπέρασαν και τα ε, όρια των όσων είχαν ε, οριστεί ως στόχοι. Ως στόχοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης. Οπότε εδώ δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι Κανείς από μας δεν ήταν στην πραγματικότητα ε, αδιάφορος. Το πρόβλημα ήταν να λυθεί το θέμα του δημόσιου χρέας, χρέους. Ερωτώ λοιπόν, ποιες ήταν οι χώρες που υλοποίησαν ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις με στόχους που είχε ε, ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες είναι οι χώρες που συμμορφώθηκαν ενώ για κάποιους άλλους ε, βλέπουμε ότι τελικά το δημόσιο πολλαπλασιάστηκε και υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε πού ακριβώς ε, χρησιμεύει η νομοθεσία. Οι επενδύσεις, οι δημόσιες επενδύσεις κατέρευσαν και συνεχίζουμε να έχουμε αυτή την αιμονή την ευρωπαϊκή κατά των ε, κρατικών επενδύσεων. Βλέπουμε λοιπόν την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι μια τεράστια κοινωνική κρίση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες με πτώση του ΑΕΠ σε πολλές από τις χώρες αυτές. Ποιο είναι λοιπόν ο αντίκτυπος της νομικής ε, ενοποίησης και του policy mix που αναφέρει και η συγγήτρια. Νομίζω υποχρεούμαστε να κάνουμε τη σχετική ανάλυση. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων που ε, κάνει και η συγγήτρια, όμως είναι σημαντικό να δούμε αν τα νομοθετικά ε, πακέτα που εγκρίθηκαν μπόρεσαν να αναχαιτήσουν τα προβλήματα αυτά ή αν αντιθέτως τα επιδίνωσαν. Εγώ βλέπω και κατά την άποψή μου επιδίνωση. Δεν μπορώ να μακρηγορήσω, ξέρω ότι πρέπει να, να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά σε κάθε περίπτωση ήθελα πολύ γρήγορα να σχολιάσω και κάποια από τα σημεία που φύγει η εισηγήτρια για να προχωρήσει όλη η συζήτηση. Η εισηγήτρια αναρωτιέται εάν το πακέτο της οικονομικής διακυβέρνησης μπορεί με ε, όσα προτείνει να διασφαλίσει ένα σωστό πώληση μίξ. Εγώ πιστεύω πως όχι και δεν υπάρχει και τέτοιο τρόπος. Επίσης, η συγγήτρια αναρωτιέται αν υπάρχουν δημοσιονομικές πολιτικές στην Ευρωζώνη που να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα τα, της κυκλικής διασύνδεσης εάν υπάρχει τέτοιο δυναμικό και εγώ θα απαντούσα πως ναι, υπάρχει αλλά λείπει η κινητοποίηση. Ποιο είναι το κατάλληλο policy mix, αυτή είναι μια άλλη ερώτηση, εδώ πρέπει να απαντήσουμε, θα έλεγα αύξηση των δημόσιων κρατικών επενδύσεων και από την άλλη εγγύηση των εισοδημάτων, διότι χωρίς εγγύηση των εισοδημάτων ε, πώς θα υπάρξει ζήτηση. Μόνο η ζήτηση μπορεί να στηρίξει τη σωστή δημοσιονομική πολιτική. Επίσης, ως προς τις πολιτικές που έχουν να κάνουν για τις χώρες με τα μεγάλα ελλείμματα στην Ευρωζώνη. Εδώ θα μπορούσε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, θα μπορούσε να γίνει η στήριξη της εσωτερικής ζήτησης, αλλά όλες αυτές οι ιδέες δικαίως αναφέρονται αλλά εάν υπήρχε στήριξη της συνολική ζήτησης, τα προβλήματα αυτά θα είχαν απαντηθεί και θα υποφελούνταν ιδίως οι χώρες που έχουν τα προβλήματα ελλείμματος ως προς την ευελιξία και εδώ δεύω προς το τέλος της παρέμβασής μου για την ευελιξία των ισχυών των κανόνων. Διερωτάται η συγκεκριμένη οικονομική διακυβέρνηση συμβάλλει ή όχι στην μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Εδώ θα έλεγα πως όχι. Όχι απλώς δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών, αλλά επιδεινώνει την κατάσταση εντός των επιμέρους κρατών και τίθεται ακόμη και το θέμα της ευελιξίας, της διαλεκτικότητας. Ε, διερωτάτε η αν πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, πιστεύω ότι προς στιγμήν εάν πρέπει να... Πριν από το ερώτημα για το αν πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι οι τωρινοί κανόνες, το πρώτο ερώτημα πρέπει να θέσουμε αν οι τωρινοί κανόνες είναι εύστοχοι ή όχι. Διαρκώς μιλάμε για ευελιξία, για μεγαλύτερη διαλλακτικότητα και τελικά δεν ερωτιόμαστε για και το λόγο ύπαρξης των κανόνων αυτών. Και ένα τελευταίο ερώτημα για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια μέτρησης του ε, ελλείμματο. Ε, το πλαίσιο του ε, Συμφώνου Ανάπτυξη και Σταθερότητα. Είναι ένα από τα βασικά ε, θέματα που τίθενται. Θα πρέπει να δούμε αν είναι σωστά ε, τα κριτήρια για τον υπολογισμό του δημόσιου ελλείμματο. Αλλά βάσει του τωρινού συστήματος, των τωρινών κριτηρίων, δεν μπορούμε να έχουμε οικονομίε με 20% διαφορετική ανεργία. Διαθωτικό έλλειμμα μάλλον. Εδώ ε, πρέπει λοιπόν ε, μέσα σε αυτές τις εύστοχες ερωτήσεις της εισηγήτριας να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Θα έχω πάρα πολλά σχόλια να κάνω και πιστεύω ότι αυτή η αξιολόγηση και αναθεώρηση είναι όχι απλώς εύστοχη αλλά απολύτως αναγκαία και επίγουσα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συνεδρίαση μας στις 12.30 οπότε θα ζητήσω τον επόμενο μιλητή να σεβαστεί τα χρονικά όρια. Τρία λεπτά το πολύ για να μπορέσει και η συγκήτρια να κάνει μια καταληκτήρια παρέμβαση. Με συγχωρείς Ελίζα. Μπορούμε όμως να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει η κυρία Φεραίρα. Σας είπα το χρονοδιάγραμμα και υπάρχει και συνάντηση ειδικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν προβλέπεται για σήμερα, ούτε υπάρχει ο χρόνος. που Σύντομος να είμαι, αλλά το θέμα είναι τέτοιο που σηκώνει συζήτηση. Ευχαριστούμε την κυρία Μπερές. Συμφωνώ με πάρα πολλά από όσα ισχυρίζεται. Αυτά που την ε, ανησυχούν για ε, τι δεν έχουμε εφαρμόσει, τι έχουμε κακώς εφαρμόσει από το πακέτο. αυτοί που ανησυχούν την αύξηση του χρέους. Ακριβώς με αυτά τα μέτρα τα πράγματα τα γίνανε χειρότερα. Όταν ε, το, η πολιτική μας ομάδα έλεγε ότι αυτοακυρώνεται κατά κάποιο τρόπο το μέτρο της εξαπλής δέσμης, ε, έτσι έγινε, έτσι, έτσι, σε τέτοιο μη ενάρετο κύκλο οδήγησε και αυτή η πολιτική αναθεώρηση του πακέτου. Έχουμε και του κανόνες, ξέρουμε ότι δεν λειτουργούν, άρα θέλουμε μεταρρύθμιση. Να, ποια προβληματική πρέπει να γίνει που είναι τόσο σημαντική. Ο κ. Μοσκοβισή ήρθε και είπε ότι είναι ανοιχτό για να αρχίσει την αλλαγή όσον αφορά τη δέσμη μέτρων. Αυτό πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα-πρώτα γιατί απέτυχε και δεύτερον γιατί τώρα δεν υπάρχει ασφαλή δικαίωση όσον αφορά την εφαρμογή όλο αυτό το πακέτο και το είπε πριν και η συγγήτρια δεν έχουμε ορισμό, τι θα πει εξαιρετικές περιστάσεις δεν υπάρχει επίσης τι θα πει severe economic downturn ε, ούτε τι θα πει διαρθρωτική ισορροπή όλα αυτά, όλα αυτά τα έχει αναλάβει ένα, μια ομάδα εργασίας, ένα group και έχει τεράστια ε, διεκριτική ευκαιρία η Επιτροπή. Τι γίνεται με την εξαπλή μέτρων. Όταν θεσπίστηκε είχαμε είχαμε το, το, το, κλάσμα πάνω από το 60% του υπερβάλλοντος χρέους, ε, υπήρχαν νομικές ε, γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν. Ας κάνει ανακοίνωση η Κομισιόν, τι πρεσβεύει, τι προτίθεται να κάνει. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί τι εννοούμε με την αναφιόρηση του νομικού θέματος. Ασύμετρη λογική χαρακτηρίζει την πολιτική αυτή. Τι γίνεται όσον αφορά το ισοζύγιο τρεκουσών πληρωμών. Τι γίνεται γιατί αλλού υπάρχει έλλειμμα, αλλού υπάρχει πλεόνασμα. Αναχώρα, δηλαδή είναι διαφορετική κατάσταση. Είναι μακροοικονομικό το θέμα. Θα πρέπει να αναζητηθεί η ισορροπία τι γίνεται με το scoreboard. Πώς το πίνακα των επιδόσεων αυτός λειτουργεί. Άλλο σημαντικό. Ζητούμε μεταρρύθμιση. Τι γίνεται με τους δείκτες, τα κριτήρια. Είπε ο κ. Μοσκοβησί ότι θέλει να έχουμε κοινωνικά κριτήρια στον πίνακα επιδόσεων όπως η φτώχεια, η ανεργία, οι δημόσιες ε, υπηρεσίες, οι κοινοφελείς, όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν νομίζω ότι η μακροοικονομική πολιτική μπορεί όλα αυτά να τα αγνοήσει. Έχουμε επιδείνωση από τη λιτότητα των κρατικών υπηρεσιών παντού. Τι γίνεται με τις ε, δημόσιες επενδύσεις, τα είπε η κυρία Μάρισα Ματίας. Να γίνει εδώ διάκριση δημόσια δαπάνη, κρατική δαπάνη που έχει κάποια απόδοση ή όχι. Δηλαδή υπάρχει ή δεν υπάρχει. Απόσβεση. Σύμφωνα τώρα υπάρχει μεγάλο έλλειμμα επενδύσεων. Είμαστε πρώτον πυλών της τέσσερι, τέταρτης ύφεσης εδώ για την Ευρώπη. Άλλο σημαντικό η προβληματική που είπε η συγγήτρια όσον αφορά το κατά πόσον θα επιτραπεί κάποια ευελιξία ούτως ώστε να μπορέσουν οι χώρες να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις. Τι είδους μεταρρυθμίσεις κοινωνικές, τι αντίκτυπο έχουν, τι εξυγένση δημιουργικών έχουμε, τι γίνεται με το χρέος. Έχουμε τον ΟΣΑ που έχει αποφανθεί σε σχέση με τις επιπτώσεις επί των μισθωτών σε σχέση με τα μέτρα τα οποία λήφθησαν ή στην ε, Ισπανία. Γιατί μισθολογικά ήταν ε, καταστροφικές συνέπειες. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις προτεραιότητες που θέλουμε να καλύψουμε με αυτά τα διπλά και εξαπλά πακέτα. Σύμφωνα με τα άλλα. Και άρα θα πρέπει να δώσουμε μάχη για να γίνει νομική εκβάθρον μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ο τελευταίος τώρα. Η Ο Φλίν. Συγγνώμη που θα πρέπει να φύγω γιατί πρέπει στο δεκάμιση να βρίσκομαι κάπου αλλού. Οπότε δίνω τη σκητάλη της Προεδρίας στον ε, παρακαθήμενο του συνάδελφο Ροζάτη. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ακούσαμε πάρα πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Ευχαριστώ τον, ε, την εισηγήτρια. Βεβαίως το έγγραφο αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. γιατί βεβαίως δημιουργήθηκε η Ευρωζώνη αλλά η δημοσιονομική πολιτική έμεινε αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και μετά μας λέει το κείμενο πως ε, ε, ε, αυτό δεν συμβιβάζεται με τις τωρινές εμπειρίες. Λες και αυτό μόνο τα, μετά από τις εμπειρίες αυτές ε, ήταν προφανές. και όμως οι ευρωσκεπτικιστές το έλεγαν από τότε ότι δεν γίνεται νομισματική ένωση με 17 διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές και τώρα από τον κύριο Ντράγκε το ξέρουμε πως δεν θέλει μόνο συντονισμό της δημοσιονομικής πολιτικής αλλά και της ε, αγοράς εργασίας ακόμα και της εκπαίδευσης. Σημαντικότερο νομίζω είναι η αναγνώριση του δημοκρατικού ελλείμματος ε, που είχαμε στην σύλληψη της Ευρωζώνης. Ε, ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη του λαού σε δημοψήφισμα και τώρα το περνάμε σε άλλο επίπεδο συντονισμού. Υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο δημοκρατικού ελλείμματος εδώ πέρα και αναρωτιέμαι πραγματικά τι γίνεται στην Ιταλία με το κίνημα των πέντε αστέρων που ζητάει δημοψήφισμα για να αποφασίσουν οι Ιταλοί αν θέλουν ε, να συμφωνήσουν σε αυτούς τους κανόνες και καταλαβαίνω από το ευρωπαϊκό επίπεδο πως υπάρχει ανάγκη συντονισμού. Οπότε πρέπει ο λαός να κρίνει και εγώ θα συνιστούσα όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης να δώσουν στους, υπόλοιπους, στους λαούς τους το δικαίωμα να λάβουν μία απόφαση. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η Ευρωζώνη να λειτουργήσει ως οικονομική οντότητα. Ε, το αν θα γίνει, θα καταλήξει με ένα ή κανένα μέλος είναι άλλο ζήτημα. Αλλά δεν έχουμε ρωτήσει τους λαούς της Ευρώπης και μέχρι να τους ρωτήσουμε ο κίνδυνο είναι ότι το ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για τις ελλείψεις των εθνικών οικονομιών. Και άμα το βλέπουμε συνεχώς το ευρωπαϊκό επίπεδο ως το επίπεδο το οποίο δημιουργεί την ανεργία των νέων ή την πτώση του επίπεδου ζωής, τότε πραγματικά ε, φυτεύουμε, ε, σπέρνουμε αν θέλετε την αυριανή διχόνοια. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να μπορέσει να κρίνει εάν θέλει να ζει ε, με αυτούς τους ε, περιορισμούς. Και νομίζω πως η καλύτερη, πιο δημοκρατική και πιο οικονομική, ε, πιο λογική από οικονομική σκοπιά λύση είναι να επιστρέψει η κάθε χώρα στο νομισμά της, το οποίο θα ανατιμάται ή θα υποτιμάται αναλόγως. Αυτή είναι η θα υποτιμαται λογος αυτη ειναι η ουσια του προβλήματος. Και μέχρι να το δούμε αυτό το ζήτημα δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος. Σας ευχαριστώ κύριο Φλίν. Τελειώσαμε με τους ομιλητές σε των πολιτικών ομάδων. Και ξαναπερνάμε στην Περβάνς Περές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να πείτε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι κρίμα στο τέλος μιας ε, συνεδρίασης να γίνεται αυτή η συζήτηση. Πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι, με συγχωρείς περβάρες. Πολύ σύντομοι γιατί ε, οι μεταφραστές διερμηνείς θα φύγουν. Ναι, να τα πω αγγλικά αν θέλετε για να τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση. Λυπούμε που έχουμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων τόσο αργά στην ε, συνεδρίασή μας είναι μία από τις βασικές αμμοδιότητες αυτής της Επιτροπής και για μένα και για τα ερχόμενα χρόνια να έχουμε μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη χρειαζόμαστε. Βεβαίως ε, όλοι όσοι μίλησαν δεν είναι πλέον. Εδώ θα τους δω διμερός, Αλλά για λόγους ευγένειας Για όσου έμειναν στο τέλο, θα κάνω μια σειρά από παρατηρήσει. Να θυμίσω ότι αυτή δεν είναι έκθεση. Είναι ένα έγγραφο εργασία. Έγγραφο εργασία με ερωτηματικά. Δεν έχω ε, ε, αντιτυπώσει ε, τίποτε καταφατικά. Απλώ έχω διαπιστώσει κάποια γεγονότα προ την οικονομική κατάσταση τη Ένωση, ω προ τι πρωτοβουλίε που έχουν αναλυθεί εκτό του σώματο αυτού ή εντό αυτού του σώματο, που ή ακόμη συζητούνται και κάποια ε, θέματα που εγείρονται. Εγώ δεν επινόησα τη συζήτηση περί ευελιξίας, όπως ε, υπονόησε ο κύριος Λούκας. Απλώς ε, χρησιμοποίησα μία λέξη που αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκείνοι μας ζήτησαν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση Um, de I think um, she, opened the, door very strongly on some of issues. Ε, υπάρχουν βεβαίως κάποια άλλα σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε ε, όπως η ανασύσταση χώρες. Δεν έχω πρόβλημα να το συζητήσουμε και για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ε, που ανέφερε ο κύριος Λούκα, ή ε, όχι, ο κύριος Τόγερ, Τόρερ, ε, είναι μια συζήτηση που ευχαρίστως θα ήθελα να την κάνουμε για να δούμε τις, ε, τους ορισμούς για το τι είναι διευθυντική μεταρρύθμιση, αλλά και το πώς αξιολογεί το αντίκτυπος ανάλογα με την κατάσταση ενός κάτω μέλους. Είναι κρίσιμη σημασία και είναι μεταξύ αυτών που θα πρέπει να δούμε με προσοχή. Άκουσα τον κύριο Λούκα να λέει ότι θα πρέπει να δούμε την κατάσταση ανάπτυξης εκτός ευρωζώνη, που ήταν πιο θετική η κατάσταση και πιο αισιόδοξη λόγω της ποσοτική χαλάρωσης. Βεβαίω θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην πιστή στην ε, θητεία που έχει αναλάβει. Αυτό πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι διαφωνώ με τον κύριο Λούκας όταν λέει ότι η δημοσιονομική αρμοδιότητα είναι κυρίως εθνική αρμοδιότητα. Αυτό αντίκειται με όσα έχουν γραφτεί από την συνθήκη ε, του Μάστερτ και μετά με το άρθρο 121 της συνθήκης και επειδή τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι οικονομικές πολιτικές τους πρέπει να είναι συντονισμένες για λόγους αμοιβαίου συμφέροντος. Δεν θέλω να μακρηγορήσω αλλά θεωρώ ότι πολλές από τις ερωτήσεις που γίνονται έχουν απαντηθεί από κάποιους από τους συναδέλφους και θα ήθελα να απαντήσω σε τρία ή τέσσερα εναπομείναντα σημεία. Το πρώτο νομίζω είναι του κυρίου Τόιρερ για το πώς το σύμφωνο σταθερότητας ε, μπορεί να είναι ένα ισότιμο πλαίσιο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το μόνο ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε. Είναι ένα από τα ερωτήματα, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα η ισοτιμία, η ισότητα. Είναι και η αποτελεσματικότητα. Ένα ζήτημα, ο καλύτερος τρόπος διεξόδου για όλη την Ένωση και την Ευρωζώνη αυτή καθεαυτή. Έχει επίσης προβληθεί το επιχείρημα ότι πολλά κρατημέλη έχουν ήδη κάνει πολλά και ότι οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν παντού. Ωστόσο, αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι οι κανόνες εφαρμόζονται και εκεί που δεν αρέσουν, ε, ίσως να το δούμε και αυτό. Και η τελευταία μου παρατήρηση για ερωτηματικά που ε, τέθηκαν ως προς την ευελιξία ή να πάμε σε απευθείας αναθεώρηση των κανόνων. Νομίζω καλό είναι να πάμε βήμα το βήμα και να δούμε πού υπάρχει περιθώριο ελιγμών, πού υπάρχει ευελιξία ε, μην ανοίξουμε τώρα άλλες πόρτες εφόσον δεν χρειάζονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω ότι θα επιτρέψει τον εαυτό της να ανοίξει τις ανάλογες πόρτες όταν υποβάλλει την έκθεσή της στις 14 Δεκεμβρίου. Ε, σε αυτή τη φάση δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ελπίζω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με όλους τους χειώδεις εισηγητές και γενικώ όλου του συναδέλφου για αυτή την κρίσιμη συζήτηση. Ε, ευχαριστούμε για αυτή την τελική παρέμβαση. Κρίμα που κάποια του χιώδει έχουν φύγει πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση. Φτάνουμε όμως στο τέλος της συνεδρίασης να σας ενημερώσω ότι έχει προβλέψει διάφορε εκδηλώσει σε σχέση με την έκθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα εργαστήριο με εξωτερικού εμπειρογνώμονε, ένα εργαστήριο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια συζήτηση στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στην Ολομέλεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια δημόσια κρόαση με υψηλού επίπεδο εμπειρογνώμονε. Δεν έχουμε ακόμα το σχετικό χρονοδιάγραμμα, αλλά θα αποφασιστεί από την Επιτροπή στο προσεκέ μέλλον. Σα ευχαριστώ Κυρίω Τη λήξη.